Alors c'est comme au théâtre, mais je n'ai pas, si, pas tapé trois coups, seulement un, mais nous allons commencer. Euh, donc bonjour à tous. Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαστε μαζί μας. Μην ξεχνάτε ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται διαδικτυακά ε, είμαστε βέβαια πολύ σοβαροί μαθητές, ε, πολύ καλοί μαθητές, οπότε κανένα πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε με την έγκριση τη μερίσιας διάταξης. Την έχετε. Δεν ξέρω μήπως ε, θέλετε κάποια τροποποίηση. Έχετε κάποιο σχόλιο για την ημερήσια διάταξη. Όχι από ό,τι φαίνεται. Την υιοθετούμε λοιπόν όπως ως έχει. Για τα πρακτικά. Οι τροποποίησει, στα πρακτικά τη 23 η και 24 η Ιουνίου θα πρέπει να ανακοινωθούν στη Γραμματεία πριν από την αυριανή μέρα στι 12 το μεσημέρι. Σημειώστε το για όλου όσους θέλουν να κάνουν ε, τις αλλαγές αυτές στα πρακτικά. Και τώρα, χωρίς να περιμένουμε περαιτέρω, γιατί ξέρω ότι γενικά το πρόγραμμα των επιτρόπων είναι πολύ φορτωμένο και επειδή έχουμε και εμείς αρκετή δουλειά στο Κοινοβούλιο και έχουμε αρκετή πίεση, ε, πίεση στην Επιτροπή μας, θέλω να δώσω πάρα αυτά το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Αλγκύρντα Σεμέτα, που θα μας παρουσιάσει ένα κείμενο σχετικά με την 100% εξέταση ε, που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, στα προϊόντα. Είχαμε προβλέψει την παρουσίαση αυτή στις 12 Ιουλίου, αλλά λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Επιτρόπου δεν μπορέσαμε να κάνουμε τότε την παρουσίαση. Σήμερα θα την κάνουμε λοιπόν. Θέλω να καλωσορίσω και τα μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού και Διεθνούς Τουρισμού καθώς και των μελών της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους προσκαλέσαμε γιατί το σκάνινγκ, η εξέταση 100% αφορά ε, το διεθνές εμπόριο και τις διατλαντικές σχέσεις. Θέλω να αφήσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο. Uh, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση ε, που μου απευθύνατε να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικές με την Αμερικανική νομοθεσία περί σάρους του 100% των εμπορευματοκιβατίων με προορισμό της ΟΠΑ. Ε, καλωσορίζω τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών της Επιτροπής σας σε αυτή τη συζήτηση. Θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας παρουσιάσω εν συντομία τις ε, προσπάθειές μας ε, να εφαρμόσουμε και να εξηγήσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας ε, της αλυσίδας τροφοδοσίας. Είναι τεχνικά τα θέματα αυτά, οπότε θα είναι δύσκολο να εξασφαλίσω την προσοχή σας, αλλά θα το προσπαθήσω. Ε, σκεφτείτε τα θρίλερ και τις ταινίες που έχετε δει. Βάλτε τον εαυτό σας ε, στην ε, θέση ενός τελωνιακού που προστατεύει την εθνική ασφάλεια των πολιτιών. Η, εξα... η ενίσχυση της ασφάλειας της ε, ε, τροφοδοσίας παγκοσμίω ε, είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικό θέμα σχέσης Ευρωπαϊκών... Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών Διακυβεύονται πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες αντιπροσωπεύουν στο διμερές εμπόριο το 31% περίπου του παγκοσμίου εμπορίου. Πέρσι οι ΗΠΑ και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντάλλαξαν περίπου παραπάνω από 360 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία αγαθών. Η εισαγωγή εμπορικών φραγμών στο διατλαντικό εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο πλήγμα στις οικονομίες μας. Κατά την άποψή μας, η νομοθεσία των ΗΠΑ που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο 2007, που απαιτεί μέχρι τον Ιούλιο 2012 το 100% των εμπορευματοκιβατίων με προορισμό τις ΗΠΑ να σαρώνονται στα ξένα λιμάνια πριν ε, φορτωθούν στα πλοία είναι ένας, ένας ενδεχόμενος τέτοιος εμπορικός φραγμός. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρωτοπόρα στον καθορισμό μιας διεθνούς θέσης σε σχέση με αυτή την απέτηση και έχει εκφράσει ανησυχίε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και των διαχειριστών των λιμανιών και του ε, επιχειρηματικού κόσμου στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Τον Απρίλιο του 2008 ε, κάναμε μια προσωρινή πρώτη ε, αξιολόγηση του αντικτύπου αυτού του μέτρου. Τη στείλαμε στην Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ και συμπεριελήφθηκε στην έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που απεστάλλει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2008. Για να υποστηρίξουμε τη θέση μας ε, με ασφαλή στοιχεία, η Κομισιόν ε, ζήτησε τρεις ε, μελέτες για το αντίκτυπο του, το 100% των εμπαρματοκιβατίων στις μεταφορές και στο εμπόριο. Η Κομισιόν εξέδωσε ένα έγγραφο των υπηρεσιών της το Φεβρουάριο 2010 με τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η απέτηση σάρωσης θα δημιουργούσε σημαντικό οικονομικό βάρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά νούμερα μόνο. Η επένδυση που θα απαιτεί το έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά λιμάνια να μπορούν να πληρούν και να σέβονται τα κριτήρια των ΗΠΑ ε, θα είναι περίπου 430-430 εκατομμύρια ευρώ. Ε, πρόσθετα ε, λειτουργικά κόστη θα ανέβαιναν στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ενώ θα έπρεπε να προσληφθούν περίπου 2.200 υπάλληλοι το κόστος να ενό ενός του από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στι ΗΠΑ θα αυξανόταν κατά 10% περίπου. Τα λιμάνια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στο νέο νόμο των ΗΠΑ θα έχαναν ένα κομμάτι τη αγορά κάτι που θα σήμαινε περισσότερη κίνηση σε άλλα λιμάνια η απέτηση του 4% ε, 100% θα δημιουργούσε απώλεια, οικονομική απώλεια περίπου 10 δισεκατομμύριων ευρώ για τις ΗΠΑ ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Αν μάλιστα την ίδια απέτηση την εφάρμοζαν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο, το συνολικό κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανερχόταν στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Η ανάλυση μας επίσης προσδιορίσε ε, σημαντικά και σαφή τεχνικά επιχειρήματα κατά του ε, μέτρου αυτού που προσπαθούν να λάβουν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, η Σάρος του 100% δεν αντιμετωπίζει τις βιολογικές και χημικές απειλές. Ε, δεν ε, αποκλείει τη δυνατότητα παρέμβασης στο φορτίο μετά τη σάρωση. εστιάζεται σε ένα τρόπο μεταφοράς, ενώ χρειάζονται λύσεις για όλους τους τύπους μεταφορών, μεταφοράς η σημερινή τεχνολογία δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την απέτηση σάρωση 100%. Για παράδειγμα, η συστηματική σκάρωση, σάρωση της, των βρωματοκιβατίων που μεταφορτώνονται είναι αδύνατη στην πράξη. Όλα αυτά τα επιχειρήματα καθιστούν σαφέ ότι αν εφαρμοστεί στην Ευρώπη, η σάρωση του 100% θα οδηγούσε ε, σε απόσπαση ε, πόρων και προσωπικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα τα οποία ε, είναι λιγότερο σημαντικά από αυτά με τα οποία ασχολούνται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να ε, εφαρμόσουμε αυτή την απέτηση. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι είναι καλύτερη μια προσέγγιση βασισμένη στην διαχείριση κινδύνου και στη διεθνή συνεργασία. Έτσι θα βελτιώσουμε την ασφάλεια της αλυσίδας τροφοδοσίας. Ε, ας ε, σας περιγράψω λίγο αυτή την πολυεπίπεδη προσέγγιση μας. Πρώτον, για κάθε φορτίο που μπαίνει ή βγαίνει ε, μια σειρά πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια θα εξετάζονται και θα ελέγχονται. Θα εφαρμόζεται αυτό το μέτρο σε όλα τα φορτία που περνούν τα, τα ευρωπαϊκά σύνορα, όχι μόνο τα εμπορευματοκιβώτια και για όλους τους τύπους των μεταφοράς. Θα ζητάμε από τους εμπορευόμενους να δίνουν στα τελωνία πληροφορίες για τα εμπορεύματά τους πριν αυτά βγουν ή μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου που προβλέπεται από την τροποποίηση ασφαλείας του τελωνικού κώδικα έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Με αυτό το σύστημα ε, θα γίνεται μια συστηματική ανάλυση δεδομένων που θα επιτρέψει στα τελωνία να ελέγχουν όλα τα φορτία για να εντοπιστούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, οι οποίοι θα ελεγχθούν αργότερα. Δεύτερο επίπεδο προέρχεται από την, ε, τον εντοπισμό και την πιστοποίηση αξιόπιστων ε, οικονομικών φορέων ε, που έχουν αποδείξει και την οτροπία τους αλλά και σε πράξη την προσήλωσή τους σε θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και το πρόγραμμα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και περιλαμβάνει πάνω από 5.500 εταιρείε οι οποίες έχουν ζητήσει πιστοποίηση μεταξύ των αυτών 2.500 έχουν ήδη ήδη λάβει πιστοποίηση για λόγους ασφαλείας. Το τρίτο επίπεδο είναι η χρήση διάφορων σύγχρονων τεχνολογιών που επιτρέπουν στα τελωνία να εξετάζουν ταχύτατα ένα επαρκές ποσοστό των ε, εμπορικών ροών χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα στο νόμιμο εμπόριο. Ε, μια σειρά συσκευών ανείχνευσης ή σάρωσης με ακτίνες χρησιμοποιούνται ε, είτε εξωτερικά είτε ενσωματωμένες στα ίδια τα εμπορευματοκιβώτια. Η με ακτινες χρησιμοποιουνται ειτε εξωτερικα τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση της ε, διατήρησης ακεραιότητας του φορτίου και του εμπορευματοκιβατίου σε όλο τον κύκλο μεταφοράς. Σφράγιση, παρακολούθηση, χνηλάτιση, υιοθεσία, και σάρωση. Η Κομισιόν έχει ε, φέρει σε πέραση μια σειρά πιλωτικών προγραμμάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων, τεχνολογίας έξυπνων κουτιών, ανταλλαγής πληροφοριών και με τρίτες χώρες όπως η Κίνα. Τέτοιου είδους project είναι σημαντικά για να προωθήσουμε την τεχνολογική καινοτομία και να βελτιώσουμε την ασφάλεια παγκοσμίω. Το τελευταίο επίπεδο προέρχεται από τη διεθνή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Συνεργασία με τους διεθνείς εμπορικούς μας εταίρους προκειμένου να εντοπιστούν πιο αποτελεσματικά οι κίνδυνοι. Καλύτερες πληροφορίες, συλλογή πληροφοριών και διαμοιρασμός τους ε, μεταξύ των τελωνιακών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο θα βελτιώσει τη διαχείριση κινδύνου. Ένα σημαντικό κομμάτι της διεθνούς συνεργασίας είναι η χρήση των διεθνών μέσων και ανοιχτών προτύπων που έχουμε, όπως το SAFE, πλαίσιο για, τα, για πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων. Βελτιώνουν την προβλεψιμότητα, την συνέργεια και αποφεύγουν πρόσθετα κόστη και άχθη μέσω συστημάτων που δεν είναι διαλειτουργικά. Και τέλος, αμοιβή αναγνώριση των προτύπων ασφάλειας και προγράμματα ε, εμπορικής συνεργασίας με τους βασικούς μας εμπορικούς εταίρους για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να διευκολύνουμε το εμπόριο ταυτόχρονα. Έχουμε ήδη συμφωνίε αμοιβέ αναγνώριση με την Ελβετία και την Νορβηγία και πολύ πρόσφατα καταλήξαμε σε μια συμφωνία ε, αναγνώσεις των ανα, αναγνωρισμένων κρυμμένων οικονομικών φορέων με την Ιαπωνία. Συζητάμε με τι ΗΠΑ και με την Κίνα και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα του επόμενου μήνε. Η διεύρυνση τη ε, συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην, ε, στο πεδίο της ασφάλειας της ε, αλυσίας τροφοδοσία είναι προτεραιότητα. Προσφάτως έχουν ενταθεί οι συζητήσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και την Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ για την αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων ε, CTPAT των ΗΠΑ και AEO της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν σημαντικό επίτευγμα για τις επιχειρήσεις και ε, θα συνεισέφερε στην βελτίωση της ασφάλειας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μέχρι σήμερα, τον Ιούλιο, η προθεσμία του Ιουλίου του 2012 για την εφαρμογή της, του όρου του, της άρρωσης του 100% των εμπαρβηματοκιβατίων παραμένει ως νόμος στις ΗΠΑ. Η ε, Υπουργός Υπουργό Εσωτερική Ασφάλεια, κ. Ναπολιτάνο, ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβρη ότι δεδομένων των ε, δυσκολιών στην εφαρμογή αυτού του νόμου θα προσπαθήσει να αναβληθεί η εφαρμογή του για μετά το 2012. Αυτό έτσι κι αλλιώ προβλέπεται από την νομοθεσία. Επίσης είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προτιμάει σαφώς μια προσέγγιση, ε, μια πολυεπίπεδη προσέγγιση ε, αξιολόγηση κινδύνου. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναθεωρεί την πολιτική ασφάλεια της ε, αλυσίας τροφοδοσίας και εμείς παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία πολύ στενά. Εν μεταξύ, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ακούγονται διάφορες απόψεις ε, για το μέλλον αυτής της νομοθεσία και το πώς θα μπορούσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Δύο συνενετικές προτάσεις ε, για ε, νομοσχέδια έχουν εισαχθεί στο, στη γερουσία των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα από αυτά τα νομοσχέδια θα τροποποιούσε την απέτηση σάρωσης διατηρώντας την μάλλον εντέλλοντας τα ξένα λιμάνια να υποβάλουν τα εμπορευματοκιβώτια είτε σε ανείχνευση μέσω ακτίνων είτε σε μη παρεμβατική απεικόνηση. Όχι και στα δύο όπως τώρα. Ε, και επίσης ε, το νομοσχέδιο αυτό αναβάλει την εφαρμογή για μετά το για, για, για το 2015. Το άλλο νομοσχέδιο θα επέτρεπε την αντικατάσταση της απέτηση σάρους 100% μέσω, μια, μέσω της χρήσης ε, μέσων ε, αξιολόγησης κινδύνου. Ε, αυτά τα μέσα συμπεριλαμβάνουν το πρόγραμμα CTPAT, το CSI, το, την πρωτοβουλία δηλαδή ασφάλειας των εμπορματοκιβατίων μέσω της οποίας 58 μάλλον ε, Αμερικάνοι τελωνιακοί θα ε, εδρεύουν σε 58 ξένα ξένα λιμάνια και θα βοηθάνε στον εντοπισμό των ελέγχων, καθώς επίσης και άλλου είδους μέσα, τα οποία ήδη υπάρχουν. Αν εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους, θα, αυτό θα επέτρεπε το, αυτό που το νομοθέτημα αποκαλεί ε, έλεγχο 100%. Αυτό άλλωστε είναι και σε... Ε, συμφωνεί και συνάδει και με την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ε, χρειάζεται ε, δράση και από, και από την Βουλή και από τη Γερουσία. Στην Βουλή η υποστήριξη του, της άρρωσης του 100% ήταν ισχυρότερη, αλλά ε, και, και το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι αρκετά ευαίσθητο. Πολλοί όμως δημοκρατικοί ηγέτες έχουν γράψει στην, ε, στο Υπουργείο Εσωτερική ασφάλεια για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για το το θέμα δεν προχωράει γρήγορα. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το πού θα καταλήξει αυτή η δημοκρατική ε, νομοθετική διαδικασία και ίσως και επικίνδυνο. Ελπίζω μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο θα έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας το 2011 για μια αναθεώρηση της νομοθεσίας σάρωση. Κυρίες και κύριοι, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σάρωση του 100% των ε, έχει κερδίσει <clears throat> την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιριών, των διαχειριστών λιμανιών και των κρατών μελών ε, και την υποστήριξη <clears throat> όλου του κόσμου συμπεριλαμβανομένου και του Παγκοσμίου Οργανισμού Τελωνίων. Η Κομισιόν είναι σε τακτικέ επαφέ με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκφράζοντα τι ανησυχίε μα για την νομοθεσία και προωθώντας ε, μια εναλλακτική προσέγγιση της ασφάλειας. Το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο ε, ήταν ένα πολύ χρήσιμο φόρουμ για, τις ε, ανταλλαγές, σε αυτό τον τομέα. Θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, ελπίζω και στην επόμενη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου που θα λάβει η χώρα σε δύο μήνες περίπου στην Ουάσιγκτον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει ε, το ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία μέσω πολιτικών ψηφισμάτων και τακτικών επαφών με το Κογκρέσο των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένου και στο πλαισίου του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου. Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι παρεμβάσεις ε, έχουν αυξήσει την ε, συνειδητοποίηση στο Κογκρέσο ότι υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και ε, το Κογκρέσο έχει πλέον αντιληφθεί ότι υπάρχει και εναλλακτική προσέγγιση. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να πιέζουμε για αλλαγή στην νομοθεσία. Η προσπάθεια σας ε, με τους ομολόγους σας, ενώπιον των ομολόγων σας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ε, είναι πολύ χρήσιμες. Θα σας ε, ενημερώνουμε τακτικά για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας παρόλη την τεχνική φύση του θέματος. Ευχαριστώ. I'm Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, πλήρη παρουσίαση. Παρότι είναι τεχνικό το θέμα, είναι και εξόχως πολιτικό, γιατί η συνεργασία για τις συναλλαγές με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, όταν ε, βελτιώνεται η ασφάλεια και προωθείται η αξιολόγηση του κινδύνου, είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωφέλιμο και για τις δύο υπήρους. Θα, αφήσω τώρα το λόγο στους συντονιστές, οι οποίοι έχουν σίγουρα ερωτήσεις να σας θέσουν. Ο κύριος Σουάπς, δεν ξέρω αν έχει ερωτήσεις. Βάπς, μάλλον. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που ασχολείστε ενεργά με αυτό το θέμα. Ήδη εμείς είχαμε πει πως δεν πιστεύουμε πως ο έλεγχος 100% όλων των αγαθών είναι δυνατός τεχνικά και αν γίνεται κιόλα θα επηρεάσει πάρα πολύ το διατλαντικό εμπόριο. Γι' αυτό συμφωνώ με την άποψή σας πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, οπότε χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες σας. Δεύτερον, θέλω να υπενθυμίσω πως αυτό είναι ένα παράδειγμα για το ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς επηρεάζεται και ασχολείται όλο και πιο πολύ με αυτά τα εμπόδια του διατλαντικού εμπορίου και πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτές τις πτυχές στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα αλλά εάν μου επιτρέπετε ως τρίτο σημείο θα ήθελα να αναφέρω τον φόρο των συναλλαγών το οποίο βεβαίω υπό μια ευρύτερη έννοια μπορούμε να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε για εμένα και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, το γιατί δεν θα συνεισφέρει έστω και ένας μικρός φόρος στον ε, περιορισμό της κερδοσκοπίας. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ακούσουμε καταρχήν δύο ή τρεις ερωτήσεις και απαντάτε και στις τρεις μαζί. Η Εύλεν και Μπάρτ δεν είναι εδώ. Η Χριστέλ ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Äh, äh, Ευχαριστώ κύριε πίτροπε για, την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση που μας κάνατε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά, προφανώς. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Συμφωνώ με την Πρόεδρο και με τον Επίτροπο. Το θέμα είναι προφανώς και τεχνικό, αλλά και πολιτικό. Γιατί έχει συνέπειες στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αν φτάσουμε στη σάρωση 100%. Μας εξηγήσατε κύριε Επίτροπε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, μια και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι στο Κογκρέσο όταν ακόμα και αν αλλάζουν θέση κάποιοι, η πλειοψηφία των βουλευτών θέλουν τη σάρωση 100%. Ελπίζω λοιπόν η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε θα προσπαθήσει να επηρεάσει τα πράγματα αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει άποψη. Πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν τα πολιτικά τεκτενόμενα στο Κογκρέσο. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη, εμείς οι υπόλοιποι εταίροι των Αμερικανών δεν μπορούμε να τους στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί το θέμα δεν αφορά προφανώς την Ευρώπη όπως είπατε και εσείς αλλά και άλλους εταίρου και χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε την ανησυχία μας ε, και θα πρέπει να το κάνουμε συντονισμένα. Γιατί έχουμε εμπορικέ σχέσεις και με άλλες χώρες. Μπορούμε να συντονιστούμε λοιπόν. Διερωτώ με τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα στο Κογκρέσο ούτω ώστε να βρούμε και έναν τρόπο να το σταματήσουμε. Ο Επίτροπος θα απαντήσει στις δύο πρώτες ερωτήσεις από τους δύο πρώτους συντονιστές. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Συμφωνώ ότι παρότι το θέμα μοιάζει τεχνικό, και βεβαίως ε, για τα τελωνιακά θέματα θα πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις. Αν δούμε την ε, ευρύτερη εικόνα, το θέμα είναι και πολιτικό. Αν λάβουμε υπόψη τον όγκο ε, των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, και αν προχωρήσει αυτός ο περιορισμός θα επηρέαζε πολύ αρνητικά τις συναλλαγές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τα απαραίτητα μέτρα για να πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι η προσέγγισή τους δεν είναι η βέλτιστη. Το ερώτημά ήταν τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς από πλευράς Κομισιόν χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να πείσουμε τους Αμερικανούς να αλλάξουν την προσέγγιση και αντί για 100% σάρωση να έχουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα του Διεθνούς Οργανισμού Τελωνίων Γιατί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων πιστεύουν και εκεί ότι αυτή η σάρωση 100% δεν είναι η καλύτερη λύση. Φυσικά το θέμα αυτό είναι θέμα του Κογκρέσου. Και πολλά μέλη του Κογκρέσου εξακολουθούν να προτιμούν τη λύση της άρρωσης 100%. Από πλευράς Κομισιόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη συνάντηση που έχουμε για να πείσουμε, προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πείσουμε τους Αμερικανούς και το Αμερικανικό Κογκρέσο ακόμη και στα περιθώρια αυτής της ε, συνεδρίασης, στους διαδρόμους, να πούμε με διάφορους τρόπους τα επιχειρηματά μας ότι δεν είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και μια κοινοβουλευτική προσέγγιση. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και επιχειρήματα, ούτω ώστε να προχωρήσουμε σε ενδελεχείς ε, συζητήσεις με τα μέλη του Κογκρέσου. Νομίζω ότι με μια κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταφέρουμε να πείσουμε τις ΗΠΑ Πολιτείες να κάνουν πίσω και να μην περάσουν αυτή την νομοθεσία. Η άλλη ερώτηση αφορούσε ένα άλλο τμήμα του χαρτοφυλακίου μου, όχι τα τελωνιακά θέματα, αλλά το θέμα των, του φόρου στις οικονομικές συναλλαγές. Θα γνωρίζετε ότι σε 7 Σεπτεμβρίου πρόσφατα έγινε μια συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ όπου συναντήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Φαντάζομαι θα διαβάσατε την ανάλυση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόθεσή μας ήταν να παρουσιάσουμε το ζήτημα αντικειμενικά. Δεν έχουμε συγκεκριμένη θέση. Φόρος στις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές ή φόρος στις ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, οικονομικές δραστηριότητες. Αξιολογούμε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις ενός φόρου ούτω ώστε να συμφωνήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. και να προωθήσουμε μια λύση η οποία θα έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά. Αλλιώς, αν προωθήσουμε ένα φόρο, μπορεί να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις και στις συναλλαγές και στον όγκο της πίστοσης προς τις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η συζήτηση δεν έχει τελειώσει. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στην επόμενη συνάντηση, την άτυπη του ΕΚΟΦΗΜ θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου. Και θα ετοιμάσουμε και μία ανακοίνωση, ετοιμάζουμε ήδη μία ανακοίνωση για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, που θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο. Κάνουμε δουλειά και δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσόη. Μετά η κυρία Ρούλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Είναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όχι μόνο γιατί είναι ευαίσθητο και μια ευαίσθητη πτυχή στις ε, σχέσεις μας ε, με τη ΣΥΠΑ που είναι στρατηγικός εταίρος, είναι επίσης σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση και νομίζω πως ε, το να προετοιμαστούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια για μια σάρωση 100% είναι ένα βάρος που δεν το χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, αλλά υπάρχει και επιπλέον λειτουργικό κόστος. Η μελέτη την οποία παρουσιάσατε παρουσιάζει αυτό το κόστος ε, σαφέστατα και Παρ' όλα αυτά, εάν υπήρχε μια μεθοδοσία η οποία θα ήταν 100% σίγουρη, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη θυσία, αλλά επισημάνεται επίσης ε, και τα όρια που έχει η σάρωση των ε, κοντέινερ. Και οφείλω να σας συγχαρώ για το ότι προτείνετε και εναλλακτικέ λύσεις. Το ερώτημά μου τώρα είναι το εξή δεδομένο του ότι αυτό είναι ένα θέμα ευαίσθητο για τις ΗΠΑ και πρόσφατα Είχαμε βεβαίως και την επέτειο του δυσάρεστου γεγονότος αυτού στην ιστορία των ΙΠΑ και της ανθρωπότητας. Πρέπει να δούμε το ζήτημα της ασφάλειας και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να πείσουμε την Αμερικανική Γερουσία και το Κογκρέσο μαζί με άλλους εταίρους μας και τώρα βέβαιως αναφέρομαι στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και άλλες χώρες οι οποίες έχουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Είπατε λοιπόν πως ήδη συζητάτε με αυτές τις σημαντικές ε, τρίτες χώρες. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο μπορείτε να συντονίσετε την ε, δική μας θέση με αυτές τις χώρες. Κυρία Ρούλε, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο λάβαμε και γραπτός κάποιες πληροφορίες πριν από την ε, συνάντηση καθώς βεβαίως ε, μας ήρθαν και επιχειρήσεις σε επαφή μαζί μας γιατί ανησυχούν για αυτές τις εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πού βλέπετε ότι μπορούμε να σας στηρίξουμε, πού θέλετε στήριξη, τι κάνει το Συμβούλιο για να σας υποστηρίξει και βεβαίω ε, και το θέμα του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν είναι απλώς ένα τεχνικό θέμα γιατί μιλάμε για τον κλάδο που προκάλεσε την κρίση ο οποίος θα πρέπει βεβαίως να υπομειστεί αναλόγως και τα βάρη αυτής της κρίσης. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μας θέτουν οι ψηφοφόροι συνεχώς. Ωραία, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ. Φαίνεται πως ο φόρος ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι το πιο αγαπητό θέμα αυτές τις ημέρες. Μπορώ να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα απαντώντας ε, στον κύριο Σβάμπ. Το βλέπουμε το θέμα. Οπότε είμαστε, έχουμε λίγο υπομονή και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ε, δουλειάς μας. Σας διαβεβαιώ πώς θα είμαι αντικειμενικός στην αξιολόγηση των ε, συνεπειών ε, των προτάσεων και οπωσδήποτε έτσι θα λάβουμε την καλύτερη απόφαση η οποία βέβαια μετά πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να καταλήξουμε στην καλύτερη λύση. Τώρα, όσον αφορά τον ε, συντονισμό με άλλες χώρες. Πρόσφατα επισκέφθηκα την Κίνα και είχαμε αυτές τις ε, συζητήσεις και το βασικό θέμα ήταν ε, το θέμα των ε, πλαστών προϊόντων και είδαμε το πώς θα επιτευχθεί κάποια πρόοδος εκεί πέρα αλλά βεβαίως συζητήσαμε και το ζήτημα της άρρωσης ε, κατά 100% και οφείλω να πω πως οι κινέζικες αρχές υποστηρίζουν την προσέγγισή μας. Ανάλογη στήριξη έχουμε και από άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους ε, της Ένωσης, οπότε δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Ανατηρηφίλιο θα έλεγα για την ε, στάση μας έναντι αυτής της άρρωσης ε, κατά 100%. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια καλή ευκαιρία, εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας ε, παγκοσμίως, να πείσουμε τις είπα να βρουν μια άλλη προσέγγιση που μπορεί να έχει και καλύτερα αποτελέσματα χωρίς ε, τόσο μεγάλο κόστος όσο η σάρωση 100%. Να επαναλάβω επίσης πως θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια όταν ε, έρχονται σε επαφή με μέλη του Κογκρέσου να φύγουν αυτό το ζήτημα και βεβαίως ε, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα και η στρατηγική μας νομίζω έτυχε θετική ε, υποδοχή ε, παγκοσμίω και μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζητήσεων με το Αμερικανικό Κογκρέσο για να του πείσουμε πω ε, η απόφαση αυτή που ελήφθη πριν από λίγα χρόνια πρέπει να αλλάξει πριν τεθεί ενισχύ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Εν συνεχεία, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Μπράντμπεν από την Επιτροπή Μεταφορών και φυσικά και αν άλλοι βουλευτέ από άλλε επιτροπέ θέλουν να πάρουν το λόγο, προφανώ μπορούν να σηκώσουν το χέρι. Κάθριν. Ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρω και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και η παρουσία σας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, αυτή η άτυπη παρουσία. Καταλαβαίνω ότι αυτό το μέτρο θα έχει κόστος και δεν ξέρω αν θα έχει καθόλου ωφέλη από πλευράς ασφάλειας. Το γεγονός ότι αρέσει στα μέλη του Κογκρέσου εισάρρωση τα 100% ε, ίσως σχετίζεται με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ποιο είναι το κόστος. Ξέρω ότι στις ΗΠΑ Πολιτείες τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ε, δεν νομίζω ότι συμφωνούν όλα τα μέλη του Κογκρέσου. Συζητείτε το θέμα. Γιατί θα υπάρξει κόστος και στα αμερικανικά λιμάνια. Ε, κόστος το οποίο θα μπορούσε και χρήματα τα οποία θα μπορούσε να πάει για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία ή άλλα προβλήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξέρουμε αυτά τα στοιχεία όταν μιλάμε στου Αμερικανού. Μιλάτε για μια συντονισμένη επίση προσέγγιση. Ο πρόεδρο τη Κομισιόν θα πάει σύντομα στι ΗΠΑ. Θα θέσει αυτό το θέμα στου Αμερικανού ομολόγου του αν πάει στη Νέα Υόρκη. Και καλό θα ήταν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συναντούνται με Αμερικανούς να θέτουν αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας το κόστος. Και πραγματικά μας ανησυχεί αυτό το θέμα. Για την αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων ασφαλείας. Ε, τώρα, σε λίγο μάλλον, θα συζητήσουμε τα θέματα τυποποίησης ε, εδώ στην Επιτροπή. Και ελπίζω ο εισηγητής να λάβει υπόψη αυτά που είπατε στην εκθεσή του. Μετά από κάτι συζητήσεις που είχα το Σαββατοκύριακο επίσης ε, με έναν άλλο ευρωβουλευτή από τη Σκωτία, βουλευτή μάλλον ε, τη Σκωτία, ε, ανησυχώ για τις απώλειες θέσεις, ε, θέσεων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, δηλαδή ανθρώπους που δουλεύουν στα τελωνία. σήμερα που μιλάμε για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι συζητήσεις κάνουμε, ότι οι εργαζόμενοι στα τελωνία και που είναι η εμπροστοφυλακή της τη πρόθεσης της ασφάλειας, καταπολέμησης του εμπορίου, της εμπορίας ανθρώπων, τη της τρομοκρατίας κτλ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαφυλαχθούν οι θέσεις τους και, και να διαφυλαχθεί βέβαια και η προσπάθεια που κάνουν. Αντώνιο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ε, Επίτροπο Σεμέτα που μας παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς της ε, Κομισιόν. Χρήσιμα και αντικειμενικά αυτά τα συμπεράσματα παρόλο ε, ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελούν εικασίες. Όμως, αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε, ε, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ε, μονομέρειας στο παγκόσμιο στερεώμα της τελευταίας δεκαετίας. Οι δαπάνες εξαιτίας αυτών των μέτρων είναι τεράστια, τα τεχνολογικά μέσα δεν είναι τέλεια και τα μόνα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας ε, λύσης ε, είναι η δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας ενδεχομένως. Και ίσως και κάποια πρόοδος ε, τεχνολογική που θα είναι βέβαια αποτέλεσμα μιας τέτοιων απαιτήσεων. Όμως η στρατιωτική ιστορία αιώνων δείχνει ότι τέτοιου τύπου μηχανισμοί ελέγχου έχουν αποτύχει. Όλοι. Δεν θα δώσω Αποτε... Ε, δεν θα δώσω παραδείγματα για να μην ε, πληγώσω, να μην θίξω εθνικές ευαισθησίες, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολλά τέτοιου παραδείγματα αποτυχημένων ελέγχων τέτοιου τύπου. Αν όμως τελικά επιβάλλουν την άποψή τους οι ακραίοι ασφάλειας, μετά τις ε, εκλογές του Νοεμβρίου. Αν δηλαδή η πλειοψηφία του Κογκρέσου επιμείνει στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, έστω και λιγάκι νερωμένου, ποια είναι η δική μας αναλλακτική αντιμετώπιση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Ε, τι έχουμε στα χέρια μας μόνο όπλο την πυθό, τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, την εδραίωση μιας κοινή ε, αλληλέγγυας τάσης με τρίτες χώρες έτσι ώστε μαζί να πείσουμε και να ασκήσουμε πίεση στους ε, ε, Αμερικανούς ή μήπως ο Επίτροπος σκέφτεται και άλλες εναλλακτικές λύσεις λίγο πιο πιστικές. Ακόμα βέβαια και αν σκέφτεται δεν θα μας, ε, κάτι τέτοιο δεν θα μας αποκαλύψει ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις. Αλλά ε, εγώ ρωτάω υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Στην περίπτωση που οι εκλογές, ε, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου των ΗΠΑ μας αναγκάσουν να ακολουθήσουμε μια άλλη τακτική. Ε, δηλαδή υπάρχουν και άλλου τύπου οικονομικές πιέσεις πέραν των διπλωματικών. Ξέρω βέβαια ότι δεν μπορείτε να μου δώσετε λεπτομερή απάντηση, γιατί ακόμα και να την έχετε δεν θα μου τη δώσετε. Ευχαριστώ. Οι εναλλακτικέ λύσει έχουν πάντα τα ωριά του. Καλά κάνει πάντω και θέτει το ερώτημα. Κρόσμαν παρακαλώ τους υπόλοιπους ομιλητέ να είναι αρκετά σύντομοι, ούτω ώστε να μπορέσει ο Επίτροπος να απαντήσει και να δώσουμε και τον λόγο στα μέλη τη Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για την εικόνα που μας δώσατε. Εάν ε, οι Αμερικάνοι κάνουν αυτό το πράγμα για λόγους ασφαλείας, ε, δεν ξέρω, θα έπρεπε να δουν καλύτερα τι έγινε στην 11η Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να δείτε τι γίνεται επίση με την επιτήρηση της αγοράς. Το διαπιστώνουμε αυτό όταν γίνονται συζητήσεις, ε, γιατί μου λέ, ακούγονται στα Υπουργεία πως ε, οι διάφορες χώρες εφαρμόζουν ε, με διαφορετική ένταση, αν θέλετε, την επιτήρηση της αγοράς, αν σκεφτούμε παραδείγματος χάρη την τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αν σκεφτούμε μετά το εάν είναι εφικτό το εισάρρωση κατά 100% θα πρέπει ίσως να λάβουμε μία δέσμη μέτρων. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι προς τον κύριο Επίτροπο εάν μπορεί να μας παρουσιάσει τι προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια. Επίσης πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος και το όφελος. Εσείς τονίσατε το κόστος, αλλά φαντάζομαι πως αν υπάρχει ισχυρότερη επιτήρηση της αγοράς έχουμε ωφέλη. Σκεφτείτε εδώ πέρα την πλαστογραφία προϊόντων, προϊόντα όπως τα κινέζικα παιχνίδια και τα λοιπά, τα οποία έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά και τα οποία φτάνουν στον καταναλωτή χωρίς κανένα έλεγχο. Οπότε θα έπρεπε ίσως να σκεφτείτε ποια δέσμη, αν θέλετε, θα μπορούσαμε μέτρο να λάβουμε. Μπορεί να είναι μία ένα από αυτά η σάρωση, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες συμφωνίες έτσι ώστε να κρατάνε κάποια πράγματα ήδη στο λιμάνι και να κλείσει εκεί πέρα η μία ή η άλλη τρύπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα κύριε Επίτροπε. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως όλα τα ερωτήματα αυτά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Για το κόστος, για τις είπα οι εκτιμήσεις μας δείχνουν πως το κόστος ε, για ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως μέρος αυτού του ποσού θα το υπομισθούν και είπα. Οπότε και για αυτούς ε, έχει κόστος και από όσο ξέρω, αυτή τη στιγμή ούτε αυτοί είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα. ελαμβάνοντας υπόψη ε, το τι γίνεται στην οικονομία. Μιλήσατε επίση για το πώς θα έρθουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς στα διάφορα φόρα. Ο πρόεδρος, ο κ. Μπαρόζο, το θίγει το θέμα σε κάθε ευκαιρία και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί εμεί θεωρούμε πως ε, το να μεταβληθεί η γνώμη του Αμερικανικού Κογκρέσου είναι πολύ υψηλή προτεραιότητα. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Βεβαίω είναι απίθανο να γίνει αυτό μέχρι τις εκλογές ε, του Νοεμβρίου γιατί βεβαίως η προεκλογική περίοδος δεν προσφέρεται για ουσιαστικές αλλαγές αλλά μετά τις εκλογές νομίζω πως ε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το νέο κογκρέσο που θα προκύψει και θα προσπαθήσουμε να του πείσουμε για την ανεργία και την απασχόληση στα τελωνία είναι ένα θέμα, γνωρίζουμε πως όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ελλημάτων και χρέους και αυτή τη στιγμή εξηγιαίνουν τα δημοσιονομικά τους και λαμβάνουν μια σειρά μέτρων. Οπότε μιλάμε για μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και βεβαίω δεν εξαιρούνται και τα τελωνία και η τελωνιακή. Οπότε είναι στα χέρια των κρατών μελών να δουν ε, πώς ε, θα γίνει αυτή η εξυγένση, αλλά είμαι σε επαφή και με τους υπουργούς και προσπαθώ να τους πείσω πως ε, τα τελωνία είναι ο τομέας όπου η μείωση της απασχόλησης δεν θα εξοικονομήσει και τόσο πολλά σε σχέση με τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θα αντιμετωπίσει εάν χαλαρώσουμε τους ε, τελωνιακούς ελέγχους. Οπότε θεωρώ πως οι Υπουργοί έχουν αντιληφθεί την κατάσταση και ελπίζω να μην ε, αντιμετωπίσουν σοβαρή μείωση της απασχόλησης στα τελωνία. Για το θέμα τώρα του ποιο είναι το εναλλακτικό μας σχέδιο και ποια μέτρα θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για το μέλλον. Εμείς ελπίζουμε Έχουμε και σοβαρά επιχειρήματα για το ότι η εφαρμογή αυτού του νόμου ούτως ή άλλως ε, θα αναβληθεί. Γιατί οι πληροφορίες μας λένε πως ακόμα και η Αμερικανική διοίκηση δεν είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία από τον Ιούλιο του 2012 και αντιλαμβάνονται και αυτοί πως ε, η προσέγγιση αυτή δεν είναι η καλύτερη, κοστίζει πολύ. Και όταν ρωτήσατε για το όφελος, η δική μας η ανάλυση δείχνει πως ε, το ίδιο ή παρόμοιο όφελος ίσως και υψηλότερο μπορεί να επιτευχθεί αν εφαρμόσουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου. Γνωρίζετε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι στον τομέα αυτών μετά την ε, τροποποίηση ασφαλείας του τελωνιακού κώδικα έχουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών πρώτης αύξησης και της αναχώρησης που μας επιτρέπει να έχουμε ένα πολύ καλύτερο σύστημα πληροφοριών και βεβαίως υπάρχει και το σύστημα αυτό των εγκεκριμένων επιχειρήσεων και η άποψή μας είναι πως ε, θα πρέπει να πάμε προς μια αμοιβαία αναγνώριση των ε, συστημάτων αναγνωρισμένων επιχειρήσεων. Αυτό έχει ήδη γίνει με την Ιαπωνία και, και είχαμε και πολύ καλή πρόοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα ελπίζω να έχουμε μια συμφωνία στον τομέα αυτών. Και με το να συμφωνήσουμε βεβαίως στις εγκεκριμένες αυτές ε, επιχειρήσεις ε, θα καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να δούμε το εμπόριο με λιγότερο επικίνδυνους ε, επιτιδευματίες. Οπότε θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν ε, από μη ε, εγκεκριμένες επιχειρήσεις και μάλιστα προωθούμε τις δικές μας τελωνιακές αρχές παγκοσμίως και υπάρχει βεβαίω και το φόρουμ ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και εκμεταλλευόμαστε κάθε συνάντηση εκεί πέρα για τον σκοπό αυτόν. Οπότε θεωρώ έτσι, σε γενικές γραμμές πώς θα είμαστε έτοιμοι όποια λύση προτείνουν οι ΙΠΑ, πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε επαρκώς. Ευχαριστώ. Τώρα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, ο κ. Μπράντμπαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που επιτρέπετε και σε εμά να πάρουμε το λόγο. Έχω κάποιες ερωτήσεις και θέλω καταρχήν να πω ένα προήμιο. Ελπίζω, κύριε Επίτροπε, ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, τη ανείχνευσης, της άρρωσης των εμπορευματοκιβωτίων στις διαπραγματεύσεις, δεν θα, γίνει, δεν θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει και εσείς να συντονιστείτε, να συντονιστούν οι διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουν ενιαία και συντονισμένα στις αρχικές σας παρατηρήσεις μιλήσατε για τη σημασία των τεχνικών θεμάτων στις διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο μέσω του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου έχουν εμπλακεί σε αυτά τα θέματα, καθώς και η Επιτροπή Μεταφορών. Ε, στη Λουμπλιάνα πριν από λίγους μήνες ε, το συζητήσαμε και μάλιστα και τον Ιούνιο. Ε, συναντηθήκαμε στη Μαδρίτη με μέλη του Κογκρέσου της, ε, των ΗΠΑ και θέσαμε το θέμα. Επομένως, να μην ε, βασιστείτε μόνο στην Επιτροπή ΤΕΚ, ε, στις τεχνικές συνεδριάσεις αυτές που έχετε, γιατί και εμείς οι βουλευτές έχουμε επαφές με τα μέλη του Κογκρέσου. Τώρα, αν προωθήσουμε αυτή τη σάρωση στο βαθμό που θέλουν οι Αμερικανοί, θα υπάρξουν προβλήματα. Θα υπάρξουν προβλήματα και στη μεταφόρτωση. Από την Ευρώπη, μεταφόρτωση μέσω Καναδά, ειδικά στα, που πάνε τελικά στα βόρειο-ανατολικά και στις μεσοδυτικές πολιτείες. Παραδείγματο χάρη το λιμάνι του Χάλιφαξ. Ε, θα έχουμε τέτοια ανείχνευση ε, και στα ενδιάμεσα λιμάνια του Καναδά δηλαδή, που μετά πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπειτα, μιλήσατε για αυτά τα έξυπνα εντό αγωγικών εμπορευματοκιβώτια. Θα μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε ενδείξει ε, για το αν η Κομισιόν θέλει να προωθήσει την έρευνα για αυτά τα έξυπνα εμπορευματοκιβώτια. Ξέρω από τι συζητήσει που κάναμε στην Επιτροπή Μεταφορών ότι ακόμα είμαστε πολύ μακριά από το να φτιάξουμε την κατάλληλη τεχνολογία για να ανοιχνεύσουμε και να μετρήσουμε το βαθμό στον οποίο τα εμπορευματοκιβώτια δημιουργούν προβλήματα. Ε, και το πρόβλημα που δημιουργεί πάλι στη μεταφόρτωση. Τώρα, ένα τρίτο σημείο. Η, αν... σάρωση με ακτίνες. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Μιλάτε για παθητική ακτινοβόληση ή ενεργητική ακτινοβόληση αν μιλάμε για 100% σάρωση, υπάρχει κίνδυνος. Όπως με κάποιους σαρωτές ας πούμε, που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια, που σαρώνουν τους ε, πιβάτες. Μπορεί ας πούμε να ακτινοβολήσουμε τρόφιμα, χρησιμοποιούμε την ενεργητική ακτινοβόληση. Ελπίζω τα τρόφιμα που πηγαίνουν στην ανθρώπινη κατανάλωση να μην τα ακτινοβολούμε. Ένα τέταρτο σημείο που συνδέεται έμεσα με αυτά που είπατε αλλά που θα αποσχολεί με σίγουρο στην Κομισιόν. Πριν από κάνα δύο χρόνια και περισσότερο η Επιτροπή Μεταφορών έκανε μια πρόταση προς τον Επίτροπο Μπαγό για μια πρόταση για την ασφάλεια στην αλυσίδα τροφοδοτίας. Ε, γιατί υπήρχαν τότε κάποιες δυσκολίες και σταμάτησε η όποια δράση. Ελπίζω η οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι πρόδρομος για μια γενική πρόταση όπως αυτή που είχε προτείνει τότε ο Επίτροπος Μπαγό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις τώρα του Επιτρόπου. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και να κλείσετε και την παρουσίασή σας. Thank you uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι μάλλον τεχνικής φύσεως. Καταρχήν για τον συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθυνσίων της Κομισιόν. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι η συναδελφικότητα και ο συντονισμός είναι λέξεις κλειδιά για την Κομισιόν. Να είστε σίγουρος ότι η δική μας Γενική Διεύθυνση θα συντονίζεται και θα μιλάει πάντα με τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις εμπορίου, εσωτερικής αγοράς κλπ. Μετά και στις εισαγωγικές μου παρατήρησεις ανέφερα τον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο και είπα ότι είναι ένα από τα κανάλια που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Είναι αλήθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα κανάλια, μεταξύ αυτών και το νομοθετικό. Το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία μεταξύ νομοθετικών σωμάτων. Η παρουσίαση βάσιμων επιχειρημάτων ενώπιον του Κογκρέσου θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Τώρα για τις πιο συγκεκριμένες σας ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την, τα αγαθά που μεταφορτώνονται μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν εφαρμοστεί το σύστημα. Φαντάζομαι θα περιλαμβάνει και τη μεταφόρτωση. Και το είπα και προηγουμένως, η σάρωση κατά τη μεταφόρτωση είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολη. Από όσο ξέρω, στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο σήμερα να γίνει σε οποιοδήποτε λιμάνι. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος αυτού. Βέβαια και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο. Είναι από τα θέματα τα οποία είναι λίγο σκοτεινά αυτή τη στιγμή και πρέπει να τα συζητήσουμε με τις αρχές των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα έξυπνα εμπορευματοκιβώτια, Είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία αυτή είναι μια δύσκολη τεχνολογία στην ανάπτυξή της. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα κάποια πιλωτικά προγράμματα στο τομέα αυτό. Αλλά η ανάπτυξη τεχνολογία είναι και δαπανηρή και αργή αυτή τη στιγμή. Συνεπώς τα ΕΦΗ, e, εμπορευματοκιβώτια, είναι αντικείμενο του μέλλοντος και όχι του παρόντος. Τώρα για την ενεργετική υπαθητική ακτινοβόληση. Είναι προφανές ότι για τα τρόφιμα η ενεργητική ακτινοβόληση θα τα επιβάρνει, θα τα κατέστρεφε. Οπότε σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι ε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της αλυσίας τροφοδοσίας. Προφανώς λοιπόν αυτή η ακτινοβόληση δεν είναι η σωστή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή της παθητικής ή της ενεργητικής ακτινοβόλησης κατά περίπτωση. Μετά, για το, την παλιότερη πρόταση Μπαρό για την ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων, ε, τροφοδοσίας με τρόφιμα. η παρούσα Κομισιόν έχει υπόψη στις ε, παλιότερες προτάσεις, αλλά ε, είναι όλες υπό αναθεώρηση. Ορισμένες από τις παλιότερες προτάσεις είχαν αποσυρθεί. Ορισμένες άλλες παρέμειναν. Για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση μπαρό πρέπει να δω. Πρέπει να το δω το θέμα για να, και να το συζητήσουμε διμερώς αν θέλετε. Α, και τελικές παρατηρήσεις ε, εν συντομία. Είμαι πεπισμένος ότι το ζήτημα αυτό παρόλο ότι πολυτεχνικό είναι άκρος πολιτικό. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουν θετικά αποτελέσματα σε αυτή τη διαδικασία. Και ελπίζω ότι τα επιχείρηματά μας, και πιστεύω μάλλον ότι τα επιχείρηματά μας είναι πολύ πιστικά. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Όλα τα θέματα που θίξατε και τα θέματα της ε, Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς ε, είναι προφανώς σημαντικά τεχνικά, ε, περίπλοκα τεχνικά, αλλά και εξόχως πολιτικά. Θα ξαναβρεθούμε με όλη την Επιτροπή το 2011. Έχουμε διάφορες εργασίες για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Επομένως, στα πλαίσια της επιτροπολογίας θα ξανάρθετε για να μας δώσετε διευκρινήσει, τις οποίες χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ.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 Πολύ σύντομα, πριν τις ψηφοφορίες, οι οποίες θα είναι ούτως ή άλλως ε, σύντομες, γιατί ο κατάλογος ψηφοφοριών είναι πολύ περιορισμένος, θα ήθελα να ακούσω το λόγο, να αφήσω το λόγο στην Μπάρμπαρα Μπέιλε, που είναι η συγγήτρια για την ε, οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, για να μας εξηγήσει πολύ σύντομα τα τελευταία τεκτενόμενα επί του φακέλου αυτού ε, πριν από τον τριμερή διάλογο που θα λάβει η χώρα σήμερα το βράδυ. Αυτό ενδιαφέρει όλους μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία έτσι σύντομα να σας πω τι γίνεται μετά την ε, συνεδρία Σκορεπέρ ε, Παρασκευή πρωί και πριν τον τελευταία πιθανό συνεδρίαση απόψε γιατί νομίζω πως σύντομα θα ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Βελγική Προεδρία για τις γρήγορες ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο διάβασα εγώ στο αποτέλεσμα της Παρασκευής ήταν πολύ ικανοποιητικό για μας, για την Επιτροπή μας, για το Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να σας πω πως τα 27 κράτη-μέλη πάλεψαν ε, μέχρι το τέλος ε, για μια πολύ, για ένα πολύ πιο ευέλικτο και ευρύτατο άνοιγμα του ψηφίσματός μας, δηλαδή θέλουν να κάνουν παραθυράκια παντού οι κυβερνήσεις σε αντίθεση με εμάς που θέλουμε ξεκάθαρους και σαφείς ε, κανονισμούς χάρηκα για το ότι επιβεβαιώθηκε στην Κορεπέρ ε, η άποψή μας για ίση μεταχείριση δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων είδε το και Περιμερίας ε, θα πρέπει να μειωθούν από ό,τι φαίνεται γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποια παραχώρηση στο Συμβούλιο. Εκείνη ήθελα, εμείς θέλαμε 9%, το Συμβούλιο ήθελε 7% και βεβαίως αυτό το οποίο θα προτιμούσαν ήταν 0%. Οπότε συμφωνήσαμε στο 8% αλλά ήταν ενδιαφέρον πως πληροφορήθηκα πως ε, μπορούν με ένα κόλπο να προκύψει αυτό το 0% οπότε πρέπει να υπολογίζουμε δεν ξέρω τα πάντα. Ναι, ναι, οι Γερμανοί κύριοι εδώ πέρα χαίρονται και διασκεδάζουν γιατί ξέρουν τι εννοώ. Μετά παρέμεινε στο 60%, 60 ε, μέρες, 60 μέρες, συγγνώμη, η οροφή για τις δημόσιες επιχειρήσεις και εκεί πέρα αυτό θα χαλαρώσει με κάποιο κόλπο από ό,τι φαίνεται. Συμφωνήσαμε τουλάχιστον για τους δημόσιες φορείς και επιχειρήσεις και τον ορισμό τους. Χαίρομαι επίσης για το ότι υπάρχει εξαίρεση για τα νοσοκομεία καθώς το Συμβούλιο τώρα θα πάει στον αρχικό μας ορισμό που είχαμε συμφωνήσει στην Επιτροπή. Είχαμε, όπως ξέρετε, κυκλοφορούσαν πάλι πολύ διαφορετικοί ορισμοί Οπότε απόψε θα επανέλθουν σε αυτό το οποίο αποφάσισε εδώ η Επιτροπή μας και αυτό είναι θετικό. Επίσης ε, εκεί που έπρεπε να υποχωρήσουμε ήταν στο ότι αυτή η ρύθμιση θα είναι προαιρετική, δηλαδή μπορούν να την εφαρμόσουν τα κρατημέλη αλλά μπορούν και να μην το κάνουν. Οπότε εκεί πέρα αναμένουμε τη βοήθεια βεβαίως των εθνικών βουλευτών που θα εκτιμήσουν και ξέρουν καλύτερα την ε, πραγματικότητα εκεί πέρα, στον, σε ποιο βαθμό δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού και να ε, αποφασίσουν. Να υπενθυμίσω πως ε, υπάρχει, εδώ πέρα μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση, μπορούν να φτάσουν το επιτόκιο και στο 9% τα κράτη-μέλη αν το επιθυμούν. Εμείς στην οδηγία συμφωνήσαμε στο 8% οπότε συνολικά ικανοποιητικά τα πράγματα. Το ικανοποιητικό αυτό αποτέλεσμα προέκυψε απόψε από ό,τι φαίνεται που θα είναι η τελευταία συνάντηση προέκυψε γιατί το Κοινοβούλιο εμφανίστηκε ενωμένο στις διαπραγματεύσεις κάτι το οποίο δεν έκανε το Συμβούλιο υπήρχαν εκεί πέρα διάφορα συμφέροντα και εμείς οι βουλευτές ε, Είχαμε βεβαίω και ομόφωνη απόφαση στην Επιτροπή μα, αλλά και εκεί πέρα στι διαπραγματεύσεις εμφανιστήκαμε ενωμένοι. Οπότε ευχαριστώ και τους σκιώδεις ηγητές εδώ πέρα και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα, που τονίζεις ότι εν τη ενώση ισχύει και από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά έχουμε την συναπόφαση πιο γενικευμένη. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανες. Ευχαριστούμε και όλους τους σκιώδεις ηγητές. Θα τα ξαναπούμε σήμερα το βράδυ στον τριμερή διάλογο. Φυσικά σε μια επόμενη συνεδρίαση θα ενημερωθείτε συνάδελφοι. Ε, θα πάμε τώρα στις ψηφοφορίες και σε 10 λεπτά θα πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω μια άλλη συνεδρίαση σε μια άλλη επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με την έκθεση Μπουσόη. Κύριε Μπουσόη, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία με συμβαστικές τροπολογίες που είναι ίδιες με αυτές της γνωμοδότησης ε, Παντσέρη για, τις για τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ και τους κοιόδης προφανώς συζητητές αλλά και τον εκπρόσωπο της Γραμματείας. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Δεν χρειάζονται κάρτες νομίζω. Ούτως ή δεν νομίζω ότι τις έχετε όλοι μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Παράγραφος 2. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. κατά αποχές 34 ψήφοι κατά σαφές παράφος 2 δεύτερη τροπολογία υπέρ κατά Αποχές. πολύ σαφές εγκρίνεται παράφος 3 τρίτη τροπολογία υπέρ Αποχέ. αποχές περνάει με αντιπλειοψηφία παράγραφος 3 β τέταρτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 σε πέμπτη τροπολογία υπέρ κατά εποχές ε, περνάει άνετα Παράφος 4 Έκτοπολογία υπερ υπέρ κατά διαθετείτε. Παράφος Παράγραφος 4α. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4β, τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, περνάει άνετα. Παράγραφος 6, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 6α. 10 τροπολογία υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 7. Εδώ είναι συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 11. Α, όχι, καταπίπτει. Παράφος 7β, 12 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράφος 8. 13 δέλτα υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο τώρα της νομοδότησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε Σουαμπ, ε, αφήνετε πάνω συνέχεια το χέρι σας, ε. Μάλλον υπέρ ήσασταν, ε, νομίζω, το ξεχάσατε το χέρι ψωμένο. 33 ψήφοι υπέρ, συγχαίρω τον εισηγητή. Τρελνόμαστε για τέτοιες ψηφοφορίες ε, εμείς οι πρόεδροι και οι γραμματείς. Σας ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία. Αλλά δεν έχω τον κατάλογο. Τον βρήκα. Θα αφήσω το λόγο στον Πιέρα Αντώνιο Παντζέρη να πει δύο-τρία προκαταρτικά λόγια πριν την ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους τους σκιώδης εισηγητές και όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτή την γνωμοδότηση. Νομίζω ότι βρήκαμε ικανοποιητικές απαντήσεις σε διάφορα σημεία και στις, στα, σημεία συμβιβασμού μέσω των προφορικών τροπολογιών. Νομίζω ότι είναι μια θετική έκθεση και θα ήθελα να την υπερψηφίσετε. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτή την γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο. Κύριε Σφαπ μπορούμε να κάνουμε μια συμπαγή ψηφοφορία, να ψηφίσουμε συλλήβδιν όλα τα σημεία. Ψηφοφορία on block. Έχει κανένα αντίρρηση για να ψηφίσουμε τουλάχιστον την πρώτη σελίδα on block. Βλέπω αντιρρήσει. Μη ένα τουλάχιστον έχει αντίρρηση. Όχι, δεν μπορούμε τότε. Έχουμε πρόβλημα μόνο με την τελευταία γραμμή, Πρόεδρε. Για μία γραμμή έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα ψηφίσουμε σημείο προς σημείο. Παράγραφος 1, πρώτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Παράγραφος 1α. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές, υιοθετείτε. Παράγραφος 2. Τρίτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Τρίτη παράγραφος. Τέταρτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 3α, η τροπολογία, υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Πάραφος 4, έκτη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Πάραφος 4, α. Έβδομη τροπολογία. Υπέρ. Υπάρχει και προφορική τροπολογία. Το κύριο Παντζέρη είναι η προφορική τροπολογία. Ο κύριο Σμιτ και ο κύριο Παντζέρη έχουν μια προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 4α, τροπολογία 7, μαζί με την Προφορική τροπολογία έχει το κείμενο δίπλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πάμε στο 4β. Το ίδιο. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία των Σμιτ και Παντζέρη. Έχει το κείμενο δίπλα στα αγγλικά. Υπέρ. κόντ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα πάλι καταπίπτει. Παράγραφος 4 γάμα. Ένα τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 5. Πρώτο συμβασμός υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Το 10 και το 11 καταπίπτει και πάμε στην πραγμα 5 5α. 12η, 12η τροπολογία υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 5β. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 6. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 15. Υπέρ. Είναι μια προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πάραφο 7. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε, Παράγραφος τροπολογία 17 στην παράγραφο 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε, Ψηφίσουμε το σύνολο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Περνάει άνετα. Συγχαρητήρια κύριε Παντζέρη. πολύ απλή, απλές οι σημερινές ψηφοφορίες. Μα ήταν πάντα έτσι. Διάλεξα καλά τη μέρα να προεδρεύσω. Σας αφήνω εγώ. Θα τα πω μια... στην επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την πειθαρχία σας. Καλησπέρα. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάμε με την έκθεση για την τυποποίηση. Ο κύριος Κουζούς Νίκ έχει το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε βεβαίω εδώ πέρα να συζητήσουμε την εσωτερική αγορά και νομίζω πως αυτό το θέμα απασχολεί συνεχώς την Επιτροπή μας, μιλάμε για την προστασία των καταναλωτών, οπότε στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρον ήταν που ακούσαμε και τον κύριο Επίτροπο γιατί ανέφερε την τυποποίηση κανένα δύο φορές. Βεβαίως σε σχέση με τις ε, διατλαντικές ε, σχέσεις και τον έλεγχο κατά 100%. Επίσης είδαμε και τις σχέσεις με Κίνα, Ινδία, οπότε είναι σαφές πως ένα παγκόσμιο πλαίσιο στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού η τυποποίηση είναι το σημαντικότερο ορόσημο που θα μας απασχολήσει και πρέπει να αναλάβουμε την ε, πρωτοβουλία. Και θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί βεβαίω μιλάμε για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα στο γενικότερο πλαίσιο της ε, Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να αναφέρω το τι έγινε τους τελευταίους 6 μήνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάλκομ Χάρμπορ, ο οποίος τα ξεκίνησε όλα αυτά. Να ευχαριστήσω και άλλους που ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδες συγκητές, ε, οι οποίοι ήταν πολύ καλή Να ευχαριστήσουμε κύριο Μπουτικόφερ από την Επιτροπή Βιομηχανίας, την Κομισιόν, γιατί βεβαίως στην αρχή η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάτι. Οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν ο Κωστής, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, μας ενημέρωσε για την τυποποίηση. Να ευχαριστήσω όλες τις οργανώσεις ε, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου, η ΣΕΝ, ΣΕΝΕΛΕΚ, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις ε, και άλλοι. Είναι λοιπόν έτοιμη η έκθεση, είναι επιτάπητος και ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πριν από 14 μέρε, όταν μεταφράστηκε η έκθεση σε όλες τις γλώσσες έχω κάποιες επιφυλάξεις για κάποιες γλωσσικές εκδοχές αλλά οπωσδήποτε θα τις εναρμονίσουμε οπότε θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία της έκθεσης η έκθεση αυτή λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτή την ε, αρχή που ισχύει ήδη. Η διτυποποίηση από ιστορική σκοπιά υπάρχει σε πάρα πολλά κρατημέλη και είναι εδρεωμένη, αλλά βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και προσπαθεί να μας δώσει μια προσέγγιση για το πώς ε, θα φύγουν αυτές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μέλων και να δούμε βεβαίω και ποιε είναι οι ομάδες των ενδιαφερομένων που συμπεριλαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, οργανώσεις που εκπροσωπούν ε, διάφορες ομάδες ε, και το περιβαλλοντικό θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ποια είναι η δική μας η προσέγγιση για τις προδιαγραφές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στην διαδικασία τυποποίηση. Πολλές οργανώσεις δεν έχουν αυτή την πρόσβαση, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι λοιπόν πολύ φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Θέλουμε να υπάρχει υποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών. Οπότε, αν υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη, αυτή αφορά την τυποποίηση των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν πως ε, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εδώ πέρα και η καινοτομία για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μιλάμε για νέες ε, τεχνολογίες, ε, για κάτι το οποίο κατευθύνει η Ισπανική Προεδρία και πάλι εδώ πέρα βέβαια πρέπει να επικεντρωθούμε στην τυποποίηση. Και αυτό τονίζω στην εκθεσή μου. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο πλανήτη. Υπάρχουν παγκοσμίες κοινοπραξίες ε, που παράγουν προδιαγραφές σε παγκοσμίο επίπεδο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης το ότι πήγαμε στην Ελβετία, επισκεφτήκαμε λοιπόν το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και εγώ προσωπικά συναντήθηκα και με προσώπους άλλων ε, κοινοπραξιών οπότε νομίζω πως η ευρωπαϊκή τυποποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια για διάφορες ευκαιρίες όπως παραδείγματο χάρη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τον ανταγωνισμό σε σχέση με μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και διάφορες άλλες χώρες ε, που προσπαθούν ε, να ενσωματώσουν τα στοιχεία αυτά της τυποποίησης ε, στο σύστημά της. Νομίζω πως η έκθεση είναι ισορροπημένη. Θα ήθελα να επαναλάβω τώρα τις ημερομηνίε, το χρονοδιάγραμμα. Πρώτα απ' όλα 10 Μαΐου οργανώσαμε μία δημόσια κρόαση με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και ήταν βεβαίω δυνατόν να την παρακολουθήσει κανείς και μέσω του διαδικτύου. Η επόμενη μετά συνεδρίαση ήταν στις 12 και 13 Ιουλίου η ιδέα προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι μέχρι αύριο 14 ε, Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχω λάβει κάποιες ε, πολύ καλές τροπολογίες και είμαι διατεθειμένος να τους συζητήσω με τους συναδέλφους. Είμαι ήδη έτοιμος να συζητήσω οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε, όπως παραδείγματος χάρη τα δικαιώματα ψηφοφοριών και βεβαίως, εντάξει μην είμαι μόνο θετικός, να αναφέρω και κάποια άλλα ζητήματα προβληματικά, τα οποία όμως ελπίζω να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τη λογική της ε, Κομισιόν, από όσο γνωρίζω θέλουν να αναβληθεί το νομοθετικό έργο μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Είναι κρίμα να περιμένουμε τόσο. Ελπίζω να τηρήσει η Κομισιόν το χρονοδιάγραμμα. Εγώ θεωρώ πως μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουμε δει όλες τις τροπολογίες και να ψηφίσουμε στην, στο Στρασβούργο την έκθεση. Τώρα, μιλώντας για τη σημασία διαφόρων οργανισμών, εγώ θα ήθελα να έχουμε μία ενιαία θέση και όχι διάφορα έγγραφα τα οποία καμιά φορά είναι κάπως έτσι επίμαχα και είναι κρίμα το ότι δεν, δεν έχουν έρθει σε επαφή μου όλοι αυτοί οι οργανισμοί, η Sense και οι έτσι οι οποίες αναμειγνύονται εκεί πέρα. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξω σε μία κοινή θέση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση. Οπότε θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ πέρα, αλλά όπως σας είπα είμαι ανοιχτό για περαιτέρω προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Θα ακούσουμε τον σκιώδη εισηγητή και ε, το κύριο Ρικό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική. Το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Συμφωνώ ότι η βάση του ισχύοντος συστήματος είναι καλή και ότι στο μέλλον το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Οι βελτιώσεις στην έκθεση ήταν πάρα πολύ καλές, πιστεύω. Να υπογραμμίσω τον ανοιχτό χαρακτήρα της διαδικασίας τυποποίησης και το πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει τη δημοκρατία. Είναι σημαντικό να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. η φωνή τους θα πρέπει να ακούγεται πιο δυνατά. Σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση δεν είναι και πολύ ρόδινη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα στα νέα κράτη-μέλη. Οι ομάδες συμφερόντων, οι ενδιαφερόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν πολύ λίγο στην διαδικασία τυποποίησης σε πολλές χώρε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω ενδεχομένω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης. Επειδή ακριβώ η, ε, η συμμετοχή των ομάδων ενδιαφερομένων είναι ισχνή, θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές θα πρέπει ε, αυτό να θεραπευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο οι προτάσει του εισηγητή είναι πολύ καλέ. Οι ευρωπαϊκέ οργανώσει θα πρέπει να παίξουν ισχυρότερο ρόλο στην διαδικασία τυποποίηση. Πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή παραγωγής, όπω την ονομάζουμε. Είναι πολύ σημαντική σε τομεί ε, δημοσίου ενδιαφέροντο. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της όροπης προσέγγισης. Ένα άλλο ζήτημα έχει σχέση με την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ιδέα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να θεωρούνται ε, ως ιδιαίτερη κατηγορία μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων είναι εξαιρετική. Πολύ συχνά δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με μεγαλύτερες εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν γέννη όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εργασία του εισηγητή. Έκανα κάποιε ελάχιστον σημασία παρατηρήσει απλώ και προτάσει τροπολογία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση γιατί αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση και αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις μας ε, στις ακροάσεις και τα ε, κρίσιμα επίσης ε, σημεία για το πώς θα πρέπει να δούμε τις εθνικές αρμοδιότητες και ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ τυποποίησης και νομοθεσίας και ρυθμιστικών αρχών και όπως σας είπαμε μας τους ε, νομοθέτες όπως σας είπα για εμένα ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούν τα περιβαλλοντικές ενώσεις ενώσεις καταναλωτών και βέβαιω και ε, η οικονομική τους στήριξη γιατί αυτό δεν γίνεται στα κράτη-μέλη. Χαιρετίζω επίσης την πρόταση που κάνατε πως ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια δεύτερη δυνατότητα και αυτό το υποστηρίζω οπότε θα μπορέσουμε να καταθέσουμε μόνο μικρές ε, τροπολογίες και νομίζω πως κατά την απόψή μου αναφέρεται πάρα πολύ λίγο το μέσο λεπικοινωνιών και πληροφορικής αλλά νομίζω κατά τα λοιπά θα είναι αρκετά καλή έκθεση και την υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος De Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση του εισηγητή που οπωσδήποτε δίνει σημασία σε όλους τους σημαντικούς οργανισμούς. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Έχω κάποιες ερωτήσεις στις ε, παραγράφους 6 έως 8 αναφέρεται στην ανάγκη τυποποίησης της υπηρεσίας ο εισηγητής. Δεν είμαι κατά, αλλά θα ήθελα να έχουμε κάποια παραδείγματα και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια παραδείγματα είτε στο διατακτικό είτε στα εκτιμώντας για το γιατί είναι τόσο σημαντικό για να το δούμε και εμείς. Παράγραφος 9 μιλάμε για τυποποίηση στην εσωτερική αγορά και λέει και θα ήθελα εγώ να μάθω εδώ πέρα ποιοι, κάποια παραδείγματα, α πούμε, ποιοι είναι αυτοί οι νέοι τομεί ε, που αναφέρει ο συγητής. Τώρα, παράγραφος 16, κάπως πιο ουσιαστικό εδώ πέρα. Αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεννόηση και βεβαίω ε, περισσότερη συμπερίληψη και των άλλων ενδιαφερομένων, αλλά μιλάει για μια συμβολική ψήφος. Ε, δεν συμφωνώ, δεν νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο ή υπάρχει ψήφος ή δεν υπάρχει. Εννοώ πραγματική. Μία άλλη επίσης ε, ιδέα που υπήρχε στην έκθεση της γραμματείας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που είναι στην παράγραφο 20 στην παράγραφο 20 λέγεται πως είναι ή ακριβό το να καταρτίζει κανείς προδιαγραφές και όμως ε, υπάρχει ένα πιλωτικό έργο όπως λέει η Γραμματεία του Κοινοβουλίου για δωρεάν προδιαγραφές ε, και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κατά πόσο γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Τέλος, στην παράγραφο 29 απευθύνεται μία έκκληση για να γίνουν ε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα παγκόσμια. Βεβαίως καλό είναι αυτό για την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά τι σημαίνει αυτό για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το αντιλαμβάνομαι τώρα όταν μιλάμε για τη ΣΥΠΑ, Κίνα, Βραζιλία, αλλά οι μικρότερες αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει και αυτές να τις σκεφτούμε νομίζω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μάνδελς δεν είναι παρόν. Ο κύριος Κρότσμαν θα τον αντικαταστήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεχνάμε πάντα προς οι προδιαγραφές προκύπτουν από τις ε, χώρες, ε, οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναμειγνύονται και βεβαίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρυθμίσει η οικονομία από μόνη της ε, και βεβαίως αυτό αφορά την Ευρώπη στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή να υπάρχουν προδιαγραφές εκείνους που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις ε, να είναι πιο αποτελεσματικές και προσπαθούμε τώρα εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε και λέμε πως ε, δεν ε, μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ το τι κάνουν οι εθνικοί οργανισμοί και πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τόσο σωστό αυτό. Δεν νομίζω πως πάντα πρέπει να διορθώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα οποία κάνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και έχω καταθέσει και κάποιες τροπολογίες. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τις ε, επιχειρήσεις ε, γιατί βεβαίως αυτό της αφορά το να είναι δηλαδή στην τελευταία λέξη πάντα της τεχνολογίας γιατί αυτό δημιουργεί προσθέμενη αξία και επιφέρει βελτιώσεις στην εσωτερική αγορά και οπωσδήποτε πρέπει να δούμε και να αναρωτηθούμε μήπως ε, τα κράτη-μέλη ε, έχουν συμφέρον υπέρ του δίκαιου ανταγωνισμού για να δούνε το τι μπορεί να γίνει με τις προδιαγραφές ΆΙΖΟ στην πλευρά της ακεραιότητας και της αμεροληψίας. Όλα αυτά είναι πτυχές τις οποίες ε, θα φροντίσω να τονίσω με τις ε, τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Εγώ ως κοιόδης εισηγητής θα πάρω τον λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά του και για το σχέδιο κειμένου, το οποίο είναι πολύ καλοφτιαγμένο και που προσπαθεί να συνθέσει, αν θέλετε, όλα τα, όλες τις απόψεις ε, για το σύστημα της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Επίσης, ε, δίνει και ένα προσανατολισμό στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύσει την πρόταση αναθεώρησης με ένα στρατηγικό κείμενο, ούτω ώστε αυτές οι προτάσεις που θα γίνουν συνεχεία και θα ψηφιστούν και στην Επιτροπή μας να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και επομένω και εφαρμόσιμες. Για μένα σημαντικά σημεία ε, είναι τα θέματα της διακυβέρνησης, του governance. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Τη διαδικασία τυποποίηση βασίζονται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, βασικές αρχές που δεν πρέπει να αλλάξουν. Παραδείγματο χάρη, αυτό που είπε ο κ. Κρότσμαν για την εθνική εκπροσώπηση και για τη διατήρηση του εθελοντικού χαρακτήρα του συστήματος. Το θέμα είναι πολύ τεχνικό και φυσικά όλοι θα πρέπει να εκφράσουν άποψή τους και οι καταναλωτές Μία ε, προσέγγιση λοιπόν ε, διαβούλευσης ε, θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. υπόψη. Έπειτα, δύο διαφορετικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί σωστά το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή να προστατευθεί ο καταναλωτής, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία ε, των απόψεων των ε, περιβαλλοντολόγων. Επίσης, η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ακούστηκε, είναι το πιο δύσκολο σημείο να επιληθεί στα θέματα τυποποίησης. Υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωριστά. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξετάσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη μία, με διαφορετικό τρόπο, και από την άλλη τους καταναλωτές. Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι πολύ γνωστό θέμα. Ε, είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και είναι ε, και η ραχοκοκαλιά της νέας αγοράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυσκολίες. Εγώ όταν μιλάω με εκπροσώπους ε, των επιχειρήσεων αυτών, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να εκπροσωπηθούν ομοιόμορφα, ενιαία αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, οι social stakeholders και αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα, γιατί θα πρέπει ε, να εξασφαλιστεί και το δημόσιο συμφέρον. Ε, και με αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα γίνουν και πιο αντιπροσωπευτικά. Θέλω επίσης αυτές οι οργανώσεις που εξασφαλίζουν και το δημόσιο συμφέρον να εκπροσωπηθούν και να έχουν... Βέβαια, ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός. Ε, ο εντοπισμός των πρωτήτων νομίζω ότι θα πρέπει να καθοριστεί από τις επιχειρήσεις. Επομένως υπάρχει εδώ ένα θέμα με την ψηφοφορία, που, το δικαίωμα ψηφοφορίας ε, για αυτές τις οργανώσεις. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα εκπροσώπησης, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Ο διαφορετικός τρόπος εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη Υπάρχουν μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά ε, ή διαφορετικές διαστάσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον, τον γεωγραφικό εντοπισμό τους και το μέγεθός τους. Δεν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι διαφορετικές η μία από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα μέσω των μελετών αντικτύπου. Εμείς σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στο θέμα της εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτή την ανάλυση να προτείνει μια δομή, ένα τρόπο και μια αναθεώρηση της τυποποίησης, ούτω ώστε να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε προς υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κονδύλια για τη χρηματοδότησή τους, γιατί είναι προσα... Ε, σημαντικές για μας, καθώς και τις ε... οργανώσεις που εκφράζουν και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον για το καλό των πολιτών. Χρηματοδότηση λοιπόν και σε αυτές τις οργανώσεις. Έπειτα, συμφωνώντας με τον εισηγητή, νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να συζητήσουμε κάποια επιμέρους ε, σημεία σε μια μεταγενέστερη φάση, που, γιατί πρέπει πρώτα να επιλύσουμε αυτά. Και τώρα τελείωσα ως ε, σκιώδης εισηγήτρια. Τρεις ε, βουλευτές θα πάρουν το λόγο τώρα. Στάιλερ, είναι ο πρώτος, δεν ξέρω αν τον πρόφερα σωστά το όνομά του, η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστούμε τον συγητή και τους και τους συγητές. Η συγητή αυτή είναι πάρα πολύ καλή, πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να δούμε πώς λειτουργούν τα, ε, οι οργανώσεις τυποποίησης στα διάφορα κράτη-μέλη και νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να ανταλλάξουμε, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, ε, για παράδειγμα με αδελφοποίηση εθνικών οργανισμών, είναι ένας απλός τρόπος. Νομίζω ότι έχουμε τέτοιους τρόπους για να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Η επιμόρφωση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική όπως το λέει και το κείμενο. Συζητώ συγγνώμη για την θόρυβο. Ε, είναι πολύ σημαντικό επίσης να υποστηρίξουμε και τις ομάδες ενδιαφερομένων. Η κυρία Κόμη το είπε και η ίδια. Και η κυρία Ρούλε είπε κάτι παρόμοιο. Μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, συνδικάτα κλπ. Εκεί η χρηματοδότηση είναι σημαντική και πρέπει να υποστηριχθούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει που θέλουν επίση να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα νομίζω ότι ε, θα πρέπει κάπω να του ενισχύσουμε γιατί αν θέλουμε να ακούγεται η φωνή των ενδιαφερομένων, να τίθεται το θέμα του ποια είναι η πιο σημαντική από αυτέ τι φωνέ, ποιοι ε, ενδιαφερόμενοι είναι οι πιο σημαντικοί. Μετά, ε, κρατικοί φορείς. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να σχολιάσει. Είναι πολύ ε, δύσκολο να συμμετάσχουν όπως και οι τοπικές αρχές. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές τοπικές αρχές, ε, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ε, που χρειάζεται να μειώσουν πάρα πολύ τον προπολογισμό τους τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό ε, και πρέπει να διατηρήσουν κάποιους, κάποιες υπηρεσίες. Οπότε η τυποποίηση πέφτει σε προτεραιότητα. Όμως ε, ε, οι τοπικές αρχές επηρεάζονται πάρα πολύ από την τυποποίηση. Για παράδειγμα, τυποποίηση στον τρόπο κατασκευής δημοσίων κτίριων. Συνεπώ οι εθνικές αρχές ε, τυποποίησης θα πρέπει να εξετάσουν πώ μπορούν να ε, βοηθήσουν και τι τοπικέ αρχέ να συμμετάσχουν. Τέλο, καινοτομία. Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσει για την καινοτομία. Νομίζω ότι η τυποποίηση έχει σχέση, σαφή σχέση με την καινοτομία. Θα πρέπει να δούμε πώ θα διατηρηθεί αυτή η σύνδεση. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας πει πώς θα λάβει υπόψη την τυποποίηση στις προτάσεις καινοτομία που θα υποβάλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουβά. Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, έχω κάποιες ανησυχίες για την έκθεσή σας. Πριν ε, ξεκινήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η τυποποίηση είναι ένα οικονομικό επιθετικό εργαλείο για την προάσπιση της Ευρώπης. Εάν το καταλάβουμε αυτό, χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Ε, είναι ένα πολεμικό εργαλείο για να υπερασπιστήσουμε, να υπερασπίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ε, θα πρέπει μέσω της ε, δικτύωσης που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο να ευνοήσουμε την Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μία ψηφοφορία, α, ψήφο, συγγνώμη, ε, στα διεθνή φόρουμ, ε, η Κίνα επίσης μία, εμείς 27. Ε, λόγω της ιστορικής μας, των ιστορικών μας καταβολών λοιπόν, μπορούμε χάρη στον τρόπο ψηφοφορίας να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Μια και το σύστημα αυτό ευνοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος αυτού μπορεί να οδηγήσει τους εταίρους μας για με μην τους πω διεθνείς οικονομικούς ανταγωνιστές, να θέσουν ε, τις βάσεις για, νέες κανόν, για νέους κανόνες αποφάσεων. Επομένως, προσοχή. Πρέπει να προχωρήσουμε με σύνεση, προσεκτικά. Γι' αυτό, κύριε Κουσούσνικ, με ανησυχούν οι προτάσεις σας. Και να εξηγηθώ καλύτερα. Θα θυμάστε θυμήσατε μάλλον τις ε, βασικές αρχές. Χαίρομαι για αυτές. Στην παράγραφο 1 λέτε ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε ριζική αλλαγή που υποσκάπτει τις θεμελιώδεις αξίες του συστήματος. Ε, για τους λόγους που σας είπα, συμφωνώ. Υπενθυμίζετε ότι οι εθνικοί εκπρόσωποι κάθε κράτους μέλου, οι διάσημες 27 ψήφοι, στην παράγραφο 13, είναι βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Συμφωνώ και εδώ. Αυτές οι βασικές αξίες μας βρίσκουν σύμφωνους. Παραδόξως όμως, στην πρότασή σας κάνετε προτάσεις που υποσκάπτουν αυτές τις βασικές αρχές. Θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Όταν προτείνετε να εισαγάγουμε μία ψηφοφορία για τις οργανώσεις ε, που εκπροσωπούν το κοινωνικό συμφέρον, ας πούμε, να έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι κατά της αρχής που υπερασπίζεστε ότι οποιαδήποτε ριζική ας πούμε αλλαγή αποδυναμώνει το σύστημα. Αν θέλουμε λοιπόν να εισαγάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετοχή της κοινωνίας και δημοκρατία, νομίζω ότι υποσκάπτουμε τα θεμέλια του συστήματος. Άλλο παράδειγμα, λέτε ότι οι εθνικοί εκπρόσωποι είναι κομβική σημασία για το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση. Ναι, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Παράλληλα, το να προτείνετε αυτέ οι οργανώσει στου ευρωπαϊκού οργανισμού να έχουν ψήφο, έστω και συμβολικού χαρακτήρα, ενώ η εθνική θέση καθορίζεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού. Του, Παγκόσμιου Οργανισμού Τυποποίησης, νομίζω ότι χαλαρώνεται και υποσκάπτει τα θεμέλια του συστήματος. Βεβαίω, πρέπει να του δώσουμε μια θέση σε αυτούς τους εταίρου. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό νομίζω ότι οδηγεί σε αποδυνάμωση του συστήματος. Και μάλιστα αυτό που κερδίζουμε δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή αυτό που κερδίζουμε με την συμμετοχή αυτών των εταίρων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και μπορούν να εκπροσωπηθούν από τους εθνικούς τους οργανισμούς ε, χωρίς όμως να τους ε, δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι καλύπτουμε έτσι τις ανάγκες τους. Η ιστορία μας έδωσε αυτό το πλεονέκτημα. Η Ευρώπη δεν έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα, ας μην το χάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν κάνω διάφορες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να ενισχύσουμε ε, αυτές τις ε, θεμελιώδεις αρχές και να διορθώσουμε κάποιες από τις ε, διατάξεις που αναφέρει ο εισηγητής και που νομίζω υποσκάπτουν, όπως σας είπα, αυτές τις αρχές και αυτό το σύστημα. Ο κύριος Βάμπ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον εξαιρετικά ανοιχτό διάλογο σε όλη τη διαδικασία και θεωρώ πως αυτό αποτελεί και πολύ καλή προϋπόθεση για την περαιτέρω διαβούλευση αυτού του θέματος. Συμφωνώ επίσης με την σχέδιση Λαρακόμη με την οποία θα καταθέσουμε από κοινού κάποιες τροπολογίες. Τέλος θεωρώ πως οπωσδήποτε έχει δίκιο ο κ. Ζιβέν όταν λέει πως πράγματι καλό είναι να εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση 27 ψήφους αλλά ενωμένοι. Οπότε πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αλλά βεβαίως νομίζω με βάση την έκθεση του κυρίου Κόσουσνικ ε, για να αλλάξουμε πιο επικοδομητικά την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα la parola. Ευχαριστώ. Σαντεμόζε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο, οι του κ. Ζουβάν με οδήγησαν να πάρω το λόγο. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Θα πρέπει το σύστημα λιγάκι να το τραγωνίσουμε. Και νομίζω ότι έχουμε και δικαίωμα. Και σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ονομάζεται Νέα Προσέγγιση υπάρχει, υφίσταται εδώ και κάποια χρόνια και σε πολιτικό επίπεδο χρειαζόμαστε κοινού κανόνες. Για παράδειγμα, σε θέματα όπως τα παιχνίδια, τα παιδικά παιχνίδια, οι οργανισμοί τυποποίησης τους καθορίζουν αυτούς τους κανόνες. Συνεπώς, δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, είναι και κοινωνικό και πολιτικό. Θα πρέπει να βρούμε μια, έναν τρόπο να καταλήξουμε σε νέες, καλύτερες ισορροπίες. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο η έκθεση είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Η κυρία Μπρίγκμαν, Διευθύντρια Ευχαριστώ. Είμαι η νέα διευθύντρια υπεύθυνη για την τυποποίηση ε, στο, στην Γενική Διεύθυνση του κ. Ταγιάννη, που είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την έκθεση του εισηγητή. Τον συγχαίρουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκληση ό,τι αφορά τους βασικούς στόχους της μελλοντικής μεταρρύθμισης στην τυποποίηση. κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Βέβαια, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Από τη δική μας πλευρά θα χρειαστεί να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε Μιλήσαμε για τα δικαιώματα ψήφου, μιλήσαμε για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή τυποποίηση στο πλαίσιο της παγκόσμιας τυποποίησης κλπ. Η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά το τι θα προτείνουμε. Και γι' αυτό το λόγο και περιμέναμε, ε, περιμένουμε ακόμα την έκθεσή σας πριν ξεκινήσουμε την αξιολόγηση αυτή. Θέλαμε να δούμε ποια είναι η γνώμη του Κοινοβουλίου. Μετά θα ξεκινήσουμε κι εμείς να σταθμίζουμε όλες τις ανακτικές λύσεις. Η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης θα σας παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατό το 2011. Τώρα θα ξεκινήσουμε την μελέτη επιπτώσεων που όπως γνωρίζετε απαιτεί οικονομική ανάλυση, λεπτομερή οικονομική ανάλυση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις τρίτες χώρες, τα αναφέρατε και εσείς και θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Ο κ. De Jong είπε, μίλησε για τις ε, ε, πτυχές που θεωρεί ότι είναι ενδιαφέρουσες. Ακούσαμε βέβαια και αντικρώμενες απόψεις. <clears throat> Θα προσπαθήσουμε στην πρότασή μας να εξασφαλίσουμε την ισορροπία προς όφελος της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε να παραμείνουμε σε επαφή με τον εισηγητή και με όλους τους ενδιαφερόμενους, τα ενδιαφερόμενα μέλη της Επιτροπής σας και περιμένουμε η έκθεση αυτή να ψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και από πλευρά μα θα, συνεργα... θα, θα, προσφέρουμε τη συνεργασία μας σε ένα τόσο τεχνικό θέμα, σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής τώρα θα μας παρουσιάσει τα τελικά του συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της τυποποίησης. Ευχαριστώ την κυρία Μπρίκμαν. Πιστεύω ότι και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με άλλες οργανώσεις θα είναι εποφελής. Σας εύχομαι καλή επιτυχία Ελπίζω να έχετε την απαραίτητη ενέργεια και εσείς και οι συναδελφοί σας, γιατί θεωρώ πως αυτή η επόμενη χρονική περίοδος θα είναι πολύ έντονη. Άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων μου και θα προσπαθήσω να τα ενσωματώσω. Εγώ δεν είμαι ανήσυχος από τα σχόλια που άκουσα. Έμαθα πολλά ακούγοντάς τα. Εγώ επισκέφθηκα φορείς τυποποίηση σε πολλές χώρες, στη Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και Πολωνία. Πήγα και σε μικρές χώρες. Επομένως, συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι για την τυποποίηση θα πρέπει να κρατήσουμε τα ωφέλη του σημερινού συστήματος και να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική του πρόοδο και να συμφωνήσουμε για το πώς θα εξασφαλιστεί. Πέρυσι τον Νοέμβριο είχαμε συμφωνήσει ότι θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης ή θα κρατήσουμε τους εθνικούς, ιδιωτικούς, εθελοντικούς φορείς τυποποίησης. Είπαμε θα σεβαστούμε όλες τις βασικές αρχές, θα εξασφαλίσουμε την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, και την προστασία όλων των ενδιαφερομένων. Αυτό, σε αυτό είχαμε καταλήξει. Δεν μιλήσαμε τότε για πανευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. Αυτή η συζήτηση έχει λήξει. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να σχολιάσω τις επιμέρους παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Φυσικά είμαι έτοιμος να συζητήσω τα διάφορα θέματα με τους συναδέλφους για τα σημεία 6, 8, 9, 16, 29 και 30. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σας και περιμένω, προσβλέπω στην ε, μελλοντική συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ που δείχνετε ανοιχτό πνεύμα για διάλογο και αντιπαράθεση και συγχαρητήρια ακόμα μια φορά για την ε, έκθεσή σας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αύριο λύγει η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα ψηφίσουμε εδώ στις 30 Σεπτεμβρίου στην ΙΜΚΟ και στην ε, Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε το κείμενο στο Στρασβούργο. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο που είναι ο αντίκτυπο της διαφήμισης, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ζουβάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συζητήσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, ε, επί της οποίας είχα την τιμή να εργαστώ. Κάποιες σημαντικές ε, προθεσμίες, τελική ημερομηνία για την ε, υποβολή τροπολογιών εδώ είναι 5 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 26 ή 27 Οκτωβρίου και θα τις παρουσιάσουμε και αν πάει καλά το πράγμα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω τη σύντομη παρουσίαση, θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν με τις παρατηρήσεις τους σε αυτό το πολύ τεχνικό θέμα και κυρίως τους κοιόδης εισηγητές. Μερικοί μάλιστα έχουν επαγγελματική εμπειρία ε, στον τομέα αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους όσους στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου και στην Κομισιόν με βοήθησαν. Καθώς και διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις μου δώσαν διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι οι αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές τομέα της διαφήμισης, όπως προσδιορίζει, ε, προσδιορίζονται από την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ιδίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ε, τεχνικές διαφήμισης. Δεν μιλάμε για τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που καλύπτονται από μια προηγούμενη οδηγία. υπήρχε κίνδυνος βέβαια να κάνω έτσι μια παρουσίαση φιλοσοφικό-κοινωνική. Προσπάθησα λοιπόν να αποφύγω αυτόν τον κίνδυνο, αυτή την παγίδα, ελπίζω να τα κατάφερα, κάνοντας πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις. Η διαφήμιση δεν είναι ο διάβολος. Ε, συχνά στις πολιτικές μας συζητήσεις ε, έτσι τον παρουσιάζουμε. Είναι ένα υποφελές εργαλείο ε, για την εσωτερική αγορά. Ε, ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την δημιουργικότητα, βοηθάει τον καταναλωτή να επιλέξει, βοηθάει την οικονομία, μειώνει τις τιμές. Με δύο λόγια, η διαφήμιση τονώνει και βοηθάει την οικονομία. Έχει πολύ θετικές πτυχές. Αντίθετα, βέβαια, η διαφήμιση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πανάκια, υπάρχει αθέμητη διαφήμιση, υπάρχει διείσδυση στην ιδιωτική σφαίρα, διείσδυση στον ε, δημόσιο χώρο, στο, στο δημόσιο βίο, επιρροή ας πούμε των καταναλωτών κτλ. Θα ήθελα πρώτα να κάνουμε μια αξιολόγηση της σημερινής νομοθεσίας ε, και τα θέματα εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές. Θα δείτε στο αιτιολογικό κάποια στοιχεία σε κάποιες παραγράφους για αυτό το θέμα, για την αξιολόγηση της οδηγίας. Είναι σημαντικό νομίζω να βρούμε έναν τρόπο για να ενδυναμώσουμε την ε, συνεργασία, για να καταπολεμήσουμε την ε, αθέμητη διαφήμιση online. Ε, προφανώς εστιάζουμε σε αυτού του τύπου τη διαφήμιση για προφανείς λόγους. Γιατί είναι καινοτόμο εργαλείο, γιατί υπάρχουν συνέχεια νέες τεχνικές, και για, σε αυτό το πρώτο σημείο για την αξιολόγηση ισχύουσα νομοθεσία θα βρείτε διάφορα θέματα ε, που μιλάνε ας πούμε, για το πόσο καλά λειτουργεί η αυτορύθμιση συνολικά, παρότι σε ορισμένες χώρες θα πρέπει ε, να δημιουργηθεί όταν δεν υπάρχει. Ε, θα πρέπει σε άλλες δεν να βελτιωθεί εκεί που χωλαίνει. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες διευκρινήσεις για τη δύσκολη σχέση μεταξύ της αυτορύθμισης και της συνέπειές της όταν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές που ξεφεύγουν, εκφεύγουν της αυτορύθμισης. Το δεύτερο τμήμα της οδηγίας, του κειμένου μάλλον ο ομιλητής, προσπαθεί να αναλύσει διάφορα προβλήματα που ε, εγείρουν η χρήση των νέων τεχνολογιών. Είναι έτσι το πιο επίκαιρο ε, στοιχείο της έκθεσης αυτής. Εδώ Άκουσα πολλές συμβουλές από συναδέλφους από το Κοινοβούλιο και από τους σκιώδεις ηγητές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Έχω διάφορα σημεία εδώ. Ε, Παραδείγματο χάρη τη στοχευμένη ας πούμε, διαφήμιση που είναι, μπορεί να γίνει συγκειμενική. Α, μιλάω για την προσωποποιημένη διαφήμιση. Δηλαδή εντοπι, πίζουμε τα γούστα σας, την ηλικία σας, ε, διαβάζουμε καμιά φορά και τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά για να δούμε τι σας ενδιαφέρει, τι σας ανησυχεί, τι σας απασχολεί και σας στέλνουμε μια συγκεκριμένη έτσι, προσωποποιημένη διαφήμιση και συμπεριφορική αναλύουμε ας πούμε τη συμπεριφορά του χρήστη. Πρέπει να βρούμε τα πολιτικά και νομοθετικά μέσα ούτως ώστε αυτές οι διαφημίσεις να μην γίνονται παρεμβατικές, ε, και να ενοχλούν την ε, ιδιωτική σφαίρα. Γι' αυτό διάφορα μέτρα εδώ τεχνικής φύσεως ε, αναφέρονται. Προφανώς δεν είναι τέλεια, γιατί είναι περιορισμένος ο κατάλογος και φυσικά κάποια πράγματα τα έχουμε ξεχάσει. Ε, προσπάθησα βέβαια να είναι όσο πιο πλήρης ο κατάλογο, όσο πιο πλήρη τα παραδείγματα. Φερρυπίν να ενθαρρύνει παραδείγματο χάρη τη συγκέντρωση παραμέτρων, προστασία του, της ιδιωτικής σφαίρας με τα υψηλότερα πρότυπα. Παραδείγματο χάρη, διαφήμιση ας πούμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Να μπορείτε κάθε φορά να αρνείστε περαιτέρω τέτοιου τύπου ε, διαφημίσεις μέσω άμεσου link. Πάντα δεν συμβαίνει. Συχνά κάνουμε copy-paste, copy-paste και βαριόμαστε να το κάνουμε. Θα μπορούμε να το κάνουμε εύκολα. Επίσης, ε, πρέπει να γίνει έτσι μια συζήτηση στην κοινωνία μας ε, για το κατά πόσο μπορούμε να, διαβάζουμε, ε, να διαβάζουν κάποιοι, πούμε, τα προσωπικά μα email. Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να διαβάσουν τα δικά μου email. Όταν διαβάζω, ας πούμε, όταν, ας πούμε, γράφω σε κάποιον, στο γείτονά μου, ας πούμε, ότι λατρεύω τις πίτσες και αμέσως μου στέλνουν μια διαφήμιση, να πάρει να φας πίτσα από εδώ, πίτσα από εκεί. Δεν μου αρέσει αυτό. Υπάρχει αυτό το σύστημα ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί, γιατί πέρα από τον εκδοτολογικό χαρακτήρα του, του email για την πίτσα, καταλαβαίνω το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό. Ε, προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Ε, καμιά φορά φτάνουμε σε επίπεδα φρίκης ε, τύπου George Orwell. Ε, εξελίσσονται ταχύτατα. Το θέμα, παραδείγματο χάρη, της πώληση ε, ενός ονόματος, ενός προϊόντος μάλλον, που βασίζεται ε, στο όνομά του. Ας πούμε, εγώ αγοράζω Ford, Citroën, Renault, Cartier. Αγοράζω αυτά τα ονόματα και τα χρησιμοποιώ. Και αυτό παραπέμπει σε ένα site που εγώ έχω επιλέξει. Εδώ πρέπει να τεθεί το θέμα της προστασίας των ονομάτων αυτής, αυτών των εμπορικών σημάτων. Επίσης υπάρχουν και κρυφή μορφή διαφήμισης, που δεν θεωρείται από την νομοθεσία διαφήμιση, αλλά είναι πραγματική διαφήμιση και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, επίσης, ε, ε τεχνικές διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ας πούμε το δίκτυα τύπου Facebook με το κουμπάκι μ' αρέσει δεν μ' αρέσει μπορεί κανείς να κάνει διαφήμιση εύκολα. Εκφεύγοντας από όλους τους κανόνες. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Τρίτο τμήμα, προστασία των ευπαθών κατηγοριών, παραδείγματος χάρη τα παιδιά ας πούμε, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν στοχοθετημένη διαφήμιση, γιατί είναι πολύ περίεργα, πολύ ανοιχτά και έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής διαφορετική από αυτή που θα έχουν όταν γίνουν ενήλικες. Επομένως, προσοχή, ίσως θα πρέπει να, να απαγορεύσουμε την στοχευμένη διαφήμιση στα παιδιά. Τέταρτο σημείο, ίσως το πιο σημαντικό αλλά και το πιο δύσκολο να εφαρμόσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να γίνουν πεφωτισμένοι σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφημίσης, να αντιμετωπίσουν έξυπνα, να καταλάβουν τι, πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα στο net, όταν χρησιμοποιείται ας πούμε η συμπεριφορική διαφήμιση, τουλάχιστον να εμφανίζεται ας πούμε όρος αυτός στη διαφήμιση αυτή. Θα τον βοηθούσε τον, θα του στέλνει πούμε καμπανάκια του χρήστη. Και μόνο και μόνο η αναφορά αυτού του ονόματος. Ήταν σύντομη αυτή η παρουσίαση, τελειώνοντας Θέλω να πω ότι είμαι ανοιχτό, είμαι διατεθειμένος να ακούσω και προτάσεις και κριτικές και προτάσεις βέβαια για τροπολογίες. Φαντάζομαι θα ακούσω θα λάβω πάρα πολλές τέτοιες και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο με τους ε, σκιώδεις συζητητές να οργανώσουμε μια συνεδρίαση εκ νέου εργασίας. Δεν είναι η πρώτη, έχουμε ήδη, ήδη κάνει διάφορες, αλλά ακόμα μία για να δούμε πού έχουμε φτάσει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, ο, κύριο, ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο εισηγητής νομίζω ότι τα κατάφερε να συνοψίσει όλα τα ζητήματα, όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Όλες οι απόψεις που είχαν ακουστεί. Θετικό είναι ότι έλαβε υπόψη του πολλές από τις ε, απόψεις που προέκυψαν στις διάφορες συναντήσεις μας. Τα σημεία στα οποία επικεντρωθήκαμε, αυτά τα έχει αναφέρει ο εισηγητής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να σταθούμε στην ιδεολογική σκέψη, ας πούμε. Υπάρχει μια παράγραφος ολόκληρη για τα προβλήματα που συνδέονται με το ίντερνετ. Πρέπει να μιλήσουμε και για τη μικρή κρυφή διαφήμιση, για την ανάγκη προστασίας ε, των καταναλωτών και στα εκτιμώντας, όχι μόνο στο ίδιο το διατακτικό του κειμένου. Εκεί που μιλάμε για τις κατηγορίες των ευπαθών πληθυσμών, μιλάμε για την ηλικία και για κάποια ελαττώματα φυσικά ή πνευματικά. Να μιλήσουμε και για κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες που καθιστούν τους καταναλωτές ε, εύπιστους απέναντι σε ορισμένες ε, διαφημίσεις. Επίσης, θα πρέπει να βάλουμε μια παράγραφο που μιλάει για την ιδιαιτερότητα κάποιων προϊόντων, παράδειγμα χάρη φάρμακα, ε, καπνό, ε, φάρμακα ειδικά που πολλούνται online, αλκοόλ και που υπάρχει νομοθεσία στην Ευρώπη. Επίσης, δύο σημαντικά σημεία θέλω να σχολιάσω στο τέλος. Το πρώτο αφορά την αυτορύθμιση και την προσφυγή στην αυτορύθμιση. Στην ε, έκθεση μιλάμε για την αυτορύθμιση του τομέα λέγοντας ότι ενσωματώνει και λαμβάνει υπόψη ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Όταν μιλάμε για το θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών στην ιδιωτική σφαίρα, δεν αρκεί να παραπέμψουμε στο soft law. Όχι. Θα πρέπει να παρέμβουμε με νομοθετικέ πολύ συγκεκριμένε πράξει, όχι μόνο με ήπια νομοθεσία. Αντί να πούμε δηλαδή ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι μειώνονται καταναλωτέ για τον τρόπο χρήση των προσωπικών του δεδομένων, εχθέω θα ήταν να βάλουμε μια σαφή νομοθεσία στην ανάγκη ρύθμιση τη ε, συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων στο ίντερνετ. Δεύτερο σημαντικό σημείο σε ό,τι αφορά την, ε, το privacy by design, την αυτόματη συλλογή ε, παραμέτρων στο ίντερνετ. Εδώ τα πρότυπα είναι ένας μηχανισμός για να αυξήσουμε τον έλεγχο και την επιλογή του καταναλωτή. Αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να ενσωματωθούν ε, στους νέους τρόπους marketing online. Θα πρέπει λοιπόν η αναφορά ε, στην πρόθεση του privacy by design να μπει στο ίδιο το διατακτικό του κειμένου και όχι μόνο στο, στην αιτιολογική σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε μεγαλύτερο βάρος του κειμένου. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις. Ε, Φυσικά θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο. Αλλά νομίζω ότι μπορείτε έτσι πολύ αποτελεσματικά να τα εντάξετε σε αυτήν την τόσο σημαντική σας έκθεση. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρόσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση Ζουβά είναι πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει ενσωματώσει αυτήν όσα έχουμε επανειλημμένως συζητήσει μεταξύ μας και ένας και ο συγητής ε, ε, ηρεμεί, χαλαρώνει όταν βλέπει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι γνώμες. Συχνά σε αυτή την επιτροπή λέμε ότι υπάρχει μια κάποια κούραση σε σχέση με την εσωτερική αγορά, ε, υπάρχει εξίσου μια κούραση και σε σχέση με τη διαφήμιση από την πλευρά του κοινού. Γιατί βέβαια είναι χρήσιμη για την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η πολλή διαφήμιση πολλέ φορέ σκοτώνει τη διαφήμιση. Για παράδειγμα, ε, είναι σαφέ ε, πια ότι χρειάζεται να μειωθούν οι διαφημιστικέ πινακίε τη πόλη και όχι να αυξηθούν. Το ενδιαφέρον λοιπόν, η σημασία μάλλον της έκθεσης αυτής είναι ότι ε, απασχολείται με την σημερινή κατάσταση. Θα ήθελα να τα συνοψίσω όλα αυτά λέγοντας το εξής. Η διαφήμιση είναι καλή, τη χρειαζόμαστε στην οικονομία. Θα πρέπει όμως να είναι ειλικρινής ε, προς τον καταναλωτή και προς τους όλους εμπορικούς και προς όλους συναλλασσόμενους. Ένας από του κινδύνου είναι ότι η διαφήμιση συχνά πλέον μεταμφιέζεται και δεν ανακοινώνεται ως διαφήμιση. Είναι η κρυφή διαφήμιση. Τρία σημεία λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτον, το είπε και ο κύριος Παντζέρη, της αυτορύθμισης το θέμα της αυτορύθμισης. Είμαι ε, θερμός οπαδός της αυτορύθμισης, ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά την ε, διαφήμιση, γιατί έχει ε, αποδείξει την αξία της αυτορύθμισης. Όμως, αυτορύθμιση δεν σημαίνει αυτοδιαχείριση, έτσι. Εκεί που υπάρχει η αυτορύθμιση σε αυτές τις χώρες, ε, υπάρχει κι άλλη μια αρχή πάνω από τους αυτορυθμιζόμενους. Η αυτορύθμιση βοηθάει οι διάφοροι επαγγελματίες σε συνεργασία με άλλους φορείς, ενδιαφέρονους κλπ, ε, να προσπαθούν να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα που εμφανίζονται, ε, μέσα όμως σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο καθορίζει ο νομοθέτης. Η αυτορύθμιση δεν γίνεται εκτός νόμου. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε λίγο περισσότερο στην εκθεσή μας ε, <clears throat> το όριο ανάμεσα στην αυτορύθμιση και τη ρύθμιση. Λέμε χρειάζεται αυτορύθμιση και χρειάζεται και συρρύθμιση, λέει η έκθεση. Θα πρέπει να πούμε όμω καλύτερα. Η συρρύθμιση χρειάζεται εκεί που η αυτορύθμιση δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει κάπως να αλλάξουμε το κείμενο. Τι σημαίνει συρρύθμιση. Συρρύθμιση είναι εκεί που οι, οι κρατικοί φορείς αποφασίζουν από κοινού με τους επαγγελματίες. Η αυτορυθμίση είναι όταν οι επαγγελματίες προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους, εξουσιοδοτημένοι από, την, ε, από το κράτος. Η αυτορύθμιση, λέει το κείμενο, ε, δεν προβλέπει κυρώσεις, δεν επιτρέπει κυρώσεις. Όχι, υπάρχουν κυρώσεις και ε, μέσω της αυτορύθμισης. Για παράδειγμα, ε, η κοινοποίηση αυτών οι οποίοι παραβαίνουν τις, τις αρχές της αυτορύθμισης. Τώρα, για την κρυφή διαφήμιση. Θα πρέπει να πούμε κάτι ε, ρητά. Είναι απαράδεκτο, κατά την άποψή μου, επιχειρήσεις να πληρώνουν εταιρείε επικοινωνίας οι οποίες ε, προσποιούνται τους καταναλωτές στέλ και στέλνουν μηνύματα σε διάφορα site ε, για να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν το α ή το β προϊόν. Εγώ θα πρότεινα αυτό, να ζητήσουμε αυτό να απαγορευτεί. Δηλαδή να μην έχει μια επιχείρηση το δικαίωμα να πληρώνει μια εταιρεία η οποία να προσποιείται ότι είναι καταναλωτής. Γιατί είναι προφανέ ότι αν εσεί μπείτε στο ίντερνετ και δείτε ότι κάποιοι άλλοι καταναλωτέ έχουν ε, θετική γνώμη για το προϊόν το οποίο ενδεχομένω σα ενδιαφέρει να αγοράσετε, λέω είναι προφανέ ότι αυτό το σύστημα μπορεί να ε, επηρεάσει την άποψή σα με ένα τρόπο τελείω παράτυπο. Πρόκειται για μια κρυφή, μεταμφιεσμένη διαφήμιση η οποία πολύ συχνά συνοδεύεται από ε, αμάβρωση ε, της φήμης άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων. Ο καταναλωτής πιστεύει ότι τα σχόλια που διαβάζει προέρχονται από ένα άλλο ειλικρινή καταναλωτή, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι κάτι τέτοιο. Τέλος. Η, συμπεριφορική διαφήμιση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Αυτό δεν, αυτά τα προβλήματα δεν προέρχονται από το ίδιο το διαφημιστικό μήνυμα, αλλά από αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα πριν το μήνυμα. Δηλαδή, τι χρησιμοποιούμε ως προσωπικά δεδομένα του ενδυνάμει κοινού μας για να περάσουμε τη διαφήμισή μας. πρέπει να καταφέρουμε όταν δίνουμε όταν κάποιος δίνει προσωπικά στοιχεία, προσωπικά δεδομένα ε, και ε, πρέπει ε, να βάλει ένα χ σε ένα κουτάκι που επιτρέπει στην εταιρεία που συλλέγει αυτά τα δεδομένα να τα κοινοποιήσει σε άλλους, αυτό το κουτάκι θα πρέπει να είναι φάνερο, να πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι προφανές έτσι ώστε ο καταναλωτής να το βλέπει και να ξέρει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Επίση, η συμπεριφορική διαφήμιση θα πρέπει να κοινοποιείται, να δημοσιεύεται ως διαφήμιση, δηλαδή να είναι φανερή διαφήμιση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα ξέρει ότι είναι διαφήμιση και δεν θα κατηγορεί γενικότερα όλα τα διαφημιστικά μηνύματα ε, τρόπον ώστε τα, τα ξερά να καίγονται μαζί με τα χλώρα. το αντίστροφο μάλλον. Ε, είναι πολύ σημαντικό η διαφήμιση να φαίνεται ως διαφήμιση, διότι με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής μπορεί να την αποκωδικοποιήσει. Ε, δεν οδηγείται σε παρανοήσεις και στρεβλώσεις. Νομίζω ότι με κάποιες τροπολογίες ε, θα μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε. Είναι πολύ σημαντικό θέμα της εκπαίδευσης. Δεν νομίζω ότι η, η, η εκπαίδευση για τη διαφήμιση είναι κάτι περίπλοκο. Απλά πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί να δώσουμε σε αυτή την εκπαίδευση ε, στα σχολεία, ε, στα, στις σχολές δημόσιας διοίκησης, ε, σχολές μέσων ενημέρωσης, συγγνώμη, να τις δώσουμε, να δώσουμε σε αυτή την εκπαίδευση το χώρο και το χρόνο που της αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι ισχυρή η κυρία Τούρνε, την οποία βεβαίω αντικαθιστώ και ήμουν από την αρχή στη συζήτηση και πρέπει να πω πως παρατηρώ πως η έκθεση αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία συζητήσαμε και αυτά τα οποία υπάρχουν σε διάφορες μελέτες και πρέπει να πω πως ειδικά οι πρακτικές προτάσεις σας και οι γενικές αναλύσεις νομίζω είναι κάτι το πολύ θετικό ότι πηγαίνουν χέρι-χέρι. Επίσης καλό είναι πως λέτε πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι παραμετρήσεις στην εσωτερική αγορά. Πολύ καλή πρόταση και η πρόταση αυτή για μια εκστρατεία ενημέρωσης, ε, διαφώτισης για το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, επίσης για την προσωπική διαφήμιση στο ίντερνετ όλα αυτά σωστά. Έχω μόνο μία αντίφαση που ανακάλυψα, που ανέφερε και η κυρία Τούν, πως λέτε στο σημείο 1 πως ε, η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, παρέχει ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο κτλ. Αλλά μετά στο σημείο 10 λέτε πως δεν καλύπτεται η κρυμμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Και βεβαίως πράγματι έχει αυτό το πρόβλημα πως προσπάθησε αυτή η οδηγία να πάει προς την πλήρη εναρμόνιση και πλέον δεν μπορούν να ξεφύγουν από εκεί τα κράτη-μέλη, το οποίο βεβαίως δημιουργεί προβλήματα όταν έχουμε νέες εξελίξεις στη διαφήμιση, στον αθέμητο ανταγωνισμό, δηλαδή πως πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά και βεβαίως είναι κάπως πιο δυσκίνητη εδώ πέρα, νομίζω υπάρχει αυτή η μικρή αντίφαση και νομίζω πως ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε κάπως την οδηγία όσον αφορά την αντιμετώπιση του αθέμη του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. De ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με όλες τις θετικές αντιδράσεις στην έκθεση. Νομίζω πως ε, Υπάρχουν πάρα πολλές καλές ε, ιδέες εδώ πέρα και σχεδόν κανένα λάθος. Παρ' όλα αυτά θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τους περιορισμούς αυτής της έκθεσης. Λέτε πως δεν θέλετε να ασχοληθείτε με την κοινωνική ψυχολογική σκοπιά των ε, διαφημίσεων και αυτό είναι κρίμα. Γιατί πέρσι είδαμε διάφορα τέτοια πράγματα. Ένα από αυτά είναι το ίντερνετ, το άλλο είναι βεβαίως ε, το τι μπορεί να γίνει με το δημόσιο χώρο. Π.χ. σε χώρους οποίους περιμένει κανείς και παλιότερα ήταν είχε την ησυχία του, τώρα αντιμετωπίζει συνεχώς οθόνες και διαφημίσεις ε, και βλέπουμε πως πηγαίνει πιο βαθιά και εισχωρεί πιο βαθιά στο υποσυνείδητο των ανθρώπων πλέον η διαφήμιση γιατί ισχωρεί παντού και καλό νομίζω θα είναι η Κομισιόν να κάνει μία έρευνα παραδείγματο χάρη για το πρώτον ε, είναι αλήθεια πως έγινε πολύ πιο διεισδυτική και πολύ πιο μαζική η διαφήμιση από το παρελθόν και δεύτερον ποια είναι πραγματικά τα κοινωνικά αποτελέσματα τέτοιου πράγματος γιατί Φαντάζομαι πως είναι απογοητευτικό για ανθρώπους που δεν έχουν τόσα λεφτά να βλέπουν συνέχεια το τι θα μπορούσαν να αγοράσουν εάν είχαν λεφτά. Δηλαδή αυτό οδηγεί και σε εντάσεις στην κοινωνία, ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει ε, νομίζω στην έκθεση και θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορούσε να κάνει κάτι να ψάξει εδώ λίγο την υπόθεση η Κομισιόν οι ευπαθείς ομάδες και ειδικά τα παιδιά. Νομίζω η έκθεση πηγαίνει σε μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση, αλλά μην περιοριστούμε μόνο στο διαδίκτυο, διαφημίσεις στα σχολεία, σε τηλεοπτικά προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά. Το βλέπουμε αυτό και στην Ολλανδία, ότι προσπαθούν βεβαίως να το μειώσουν αυτό και βεβαίως όλα αυτά τα εμπό... τα προϊόντα τα οποία προωθούνται, τα ακριβά παιχνίδια που διαφημίζονται ειδικά στα παιδιά. Εν ολίγη. μια πάρα πολύ καλή έκθεση, αλλά θέλει βεβαίω κάποια διεύρυνση αν θέλετε και νομίζω και η κυρία Ρίλου και εγώ νομίζω θα συμφωνήσουμε στο ότι η οδηγία αφενός ε, λέτε πως ε, επαρκεί, από την όλη όμως πως ε, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές. Ε, οπότε, ναι, υπάρχει εδώ μια μικρή αντίφαση και εδώ πέρα νομίζω θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση κομισιών και τέλος ένα κάπως πιο δευτερεύον σημείο, κάπου στην αρχή, στο, προάμι, στο προήμιο, στο α, αναφέρεται πως ένα από τα, προ... τα θετικά της διαφήμισης είναι πώς καταπολεμά τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Είναι πραγματικότητα αυτό. Εγώ νομίζω πως καταπολεμα τις καταχρησεις δεσποζουσα θεσεις στην αγορα ειναι πραγματικοτητα αυτο εγω νομιζω πως ειδικα οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο διαφημιστικό προϋπολογισμό και άρα έχουν ένα τεράστιο προβάδισμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτή την τεράστια διαφήμιση μια μεγάλη. Ε, κοιτάξτε, αν πράγματι μπορείτε να μου δείξετε ότι ισχύει αυτό και είναι αλήθεια, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ. Σφάμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση πρωτοβουλίας. Η επίδραση της διαφήμισης ε, στην ε, συμπεριφορά του καταναλωτή δεν είναι τόσο δεν νομίζω να την έχει επεξεργαστεί κανείς τόσο συνολικά ποτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε νομίζω πως μας βοηθάει εδώ πέρα ο συνάδελφος και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Δεύτερον, σε αντίθεση από την κυρία Ρούλα, εγώ δεν θεωρώ πως ε, το σημείο 1 είναι σε αντίφαση με άλλα σημεία της έκθεσης, γιατί βεβαίως ε, εδώ πέρα έχει η προϋπάρξη και ένα εργαστήριο που ανέφερε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι προβλήματα B2B μεταξύ επιχειρήσεων δηλαδή. Και δεν καλύπτονται αυτά ε, από αυτή την ε, οδηγία και δεν, θα, δεν οδήγησαν βεβαίως σε μείωση της ε, προστασίας των κανονιτών, εκτός εάν ε, θεωρεί η κυρία Ρούλε πως το ευρωπαϊκό επίπεδο αντιδρά χειρότερα στις αλλαγές από ότι το εθνικό επίπεδο γιατί εντάξει μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάμε για απάτες σε τοπικό επίπεδο και άλλες οι οποίες ε, διαδραματίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θεωρώ πως η Κομισιόν είναι σε θέση να εφαρμόσει το εναρμονισμένο δίκαιο και να αντιδράσει ανάλογα. Οπότε, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις εδώ πέρα βεβαίως. Ε, δεύτερον, θεωρώ πως η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την διαφήμιση πραγματικά παρουσιάζει νέες δυσκολίες ε, και προκλήσεις και θα πρέπει να συνεργαστούμε σε νεότερα με τις άλλες αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί είναι πράγματι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ σήμερα τους καταναλωτές, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, τουλάχιστον στη Γερμανία, από όσο γνωρίζω στις διακοπές, είδαμε και αυτές τις φωτογραφίες του Google, οι οποίες μας απασχόλησαν πάρα πολύ και είναι πράγματα τα οποία θα συναντάμε όλο και συχνότερα στο μέλλον. Γι' αυτό θεωρώ πως αποτελεί μια εξαίρετη βάση αυτή η έκθεση και σας ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ, Ανδρέας. Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως η έκθεσή σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είχαμε αρκετέ συζητήσεις ε, Απόψε οπωσδήποτε και εγώ είμαι κατά της διαφήμισης που απευθύνεται σε παιδιά, αλλά κάτι το οποίο προκύπτει είναι οι διαφορές που έχουμε πολιτισμικές, να μιλάμε για την ε, διαφήμιση και αυτή είναι η διαφήμιση φαντάζομαι μεταξύ της διαφήμισης και του μάρκετινγκ που είναι μια λεπτή γραμμή οπωσδήποτε γιατί βεβαίως εκεί όπου έχει δώσει την συνένεσή του ο καταναλωτής π.χ. έχει μια κάρτα πελάτη και το ξέρουν μετά η επιχείρηση το τι αγοράζει όπως έχω εγώ και αγοράζω τη γατοτροφή ας πούμε ε, είναι προφανές ότι έχω γάτα οπότε αν μετά μου κάνουν μισή λίρα έκπτωση στην επόμενη αγορά. Εντάξει, δεν νομίζω πως ε, είναι αυτό μια συμπεριφορά η οποία ε, είναι κατακριτέα, γιατί βεβαίως όπως σας είπα εγώ έχω δώσει τη συνένεσή μου και παίρνω νου τις ερωτήσεις οποίες δεν έχει δώσει κανείς την συνένεσή του το να πούμε τώρα το ότι κάπου δεν χρησιμοποιείται το μάρκετινγκ λόγω της φύσης της ευρωπαϊκής αγοράς και αυτή η μέθοδος που περιέγραψα, δηλαδή το να προσπαθούν να κρατάνε οι επιχειρήσει πιστούς στους πελάτες, έχει γίνει ο κανόνας και κάτι το οποίο πλέον θεωρείται δεδομένο. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να ρωτήσω την Κομισιόν είναι όταν μιλάμε παραδείγματο χάρη για τι λεπτέ αυτέ αποχρώσεις στη διαφήμιση, π.χ. στην οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για το παράδειγμα που θα σας δώσω. Αν αγοράσουμε λευκές συσκευέ, π.χ. ένα πλυντήριο και μας λένε πως μας δίνουν δύο έτη δωρεάν εγγύηση. Τι κάνει παρανομή η εταιρεία τότε, γιατί δεν είναι δωρεάν, γιατί είναι κάτι που τους υποχρεώνει ο νόμος. Οπότε διαφημίζουν ότι δίνουν κάτι δωρεάν ενώ είναι υποχρεωμένοι να το δώσουν. Αυτή η εταιρεία παρανομή ε, παραβιάζει την οδηγία περί των εμπορικών πρακτικών και αν ναι, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής όταν κάτι το λένε δωρεάν ενώ είναι υποχρεωτικό να το δώσουν. Αυτές οι λεπτές αποχρώσεις είναι πολύ σημαντικές. Ζούμε σε ένα νέο κόσμο, ναι, με νέα τεχνολογία κτλ. Και ας είμαστε ειλικρινείς, εάν δεν ήταν οι νέες τεχνολογίες, εταιρείε δεν θα ήξεραν τι αγοράζουμε με και αυτές τις κάρτες που μαζεύουμε πόντους. Οπότε νομίζω πως ε, ο κύριος πίσω από το Γιόγκ ε, που μίλησε για την άσχημη πτυχή, ναι, υπάρχει αυτή η κακόβουλη πτυχή αν δεν έχει συμφωνήσει κανείς, αλλά αν έχει συμφωνήσει είναι κομμάτι του κόσμου μας ε, και Βεβαίω τα πράγματα είναι άσχημα όταν δεν έχει συμφωνήσει κανεί. Αλλιώ υπάρχει ατομική επιλογή. Οπότε σα ευχαριστώ για την συζήτηση. Οπωσδήποτε εμένα με έκανε να σκεφτώ και θα ήθελα να μου πείτε με την περίπτωση αυτή του πλυντηρίου τι γίνεται. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαγκούντα. Ε, Δεν είναι παρόν. Ο κύριος Πέτερινγκ είναι εδώ. Ναι. Ευχαριστώ τον εισηγητή από πλευράς Κομισιόν για την προσπάθειά του. Και που βάζει ψηλά αυτό το σημείο στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε την επιρροή της διαφήμισης στην ε, συμπεριφορά των καταναλωτών στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών. Ε, η διαφήμιση θέτει σημαντικά ζητήματα προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας. Το θέμα είναι κατά πόσο διαφανείς αυτές οι πρακτικές. Πέρα από τη διαφήμιση του περιεχομένου, καλό είναι οι καταναλωτές να ενημερώνονται ότι υπάρχει συλλογή των δεδομένων τους. Συχνά δεν γνωρίζουν ότι λαμβάνει η χώρα συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η νομοθεσία που υπάρχει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λέει ότι θα πρέπει η τεχνολογία να είναι ουδέτερη και να χρησιμοποιεί και να γίνει τη... Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προκλήσεις ε, στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε υπόψη μας και τις προκλήσεις ε, της ε, συμπεριφορικής διαφήμισης με την μεταρρύθμιση αυτή θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Θα ήθελα να σταθώ σε συγκεκριμένα σημεία μετά τη συζήτηση που έλαβε χώρα. Έγιναν πολλές συζητήσεις και γίνονται πολλές συζητήσεις για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τη σχετική οδηγία που είναι το βασικό νομοθέτημα για την ε, διαφήμιση. Για να δούμε αν θεωρείται θεμητή ή όχι η διαφήμιση. Για την ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας αυτής, η έκθεση λέει ότι στα κράτη-μέλη ε, ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο αυτή η οδηγία και εφαρμόζεται. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν ε, λανθασμένες ενσωματώσεις ε, στην εσωτερική νομοθεσία. Εμείς το εξετάζουμε αυτό το θέμα και αν χρειαστεί θα εκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση. Η οδηγία επίτηδες είναι ευρεία και βασίζεται σε κάποιες γενικές ρήτρε. Χτίζεται γύρω από γενικές ρήτρε, ούτω ώστε να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογή. Και κάτι που είναι σημαντικό για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ε, η οδηγία αυτή ε, μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις, στις μελλοντικές προκλήσεις και να χρησιμοποιείται ε, και στο μέλλον για την καταπολέμηση των θέμετων πρακτικών και στο ίντερνετ. Το λέει αυτό η έκθεση. για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ερμηνεία, ούτω ώστε η εφαρμογή της οδηγίας να γίνει πιο ομοιόμορφη, έχουμε ε, δημοσιεύσει και κάποιες κατευθυντήρε γραμμές. Οι εθνικές ε, αρχές για την εφαρμογή το θεωρούν πολύ θετικό βήμα. Και όπως είπε ο εισηγητή, η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ε, την επικαιροποίηση αυτού του κειμένου κατευθυντηρίων γραμμών, ούτω ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τι εκάστοτε εξελίξει. Εμείς επίσης ε, αναπτύσσουμε και μια βάση δεδομένων με νομολογία και εθνικές πρακτικές που νομίζω είναι σημαντικές για τις αρχές των κρατών μελών τόσο να εφαρμόσουν και να, να ερμηνεύσουν καταρχήν και μετά να εφαρμόσουν με ενιαίο τρόπο την οδηγία. Ακούστε για ένα σημαντικό σημείο επίσης για την κρυφή διαφήμιση. Που ανέφερε και ο κ. Γοσφό. Η οδηγία, απαντώ και στην κυρία Ρούλερ, η οδηγία εφαρμόζεται και στην κρυφή διαφήμιση. Αφορά και την κρυφή διαφήμιση. Εφόσον υπάρχει μια εταιρεία πίσω από τη διαφήμιση που πλήρωσε ας πούμε καταναλωτές ας πούμε σε κάποια blog για να εκφράσουν απόψεις για διάφορα προϊόντα. Αυτό καλύπτεται από την οδηγία για τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές και θεωρείται αθέμητη πρακτική. Αυτό που δεν καλύπτεται είναι η απλή γνώμη ενός ε, μεμονωμένου καταναλωτή για το αν είναι καλό ή κακό ένα προϊόν. Τέτοιε ε, γνώμες ε, απλώνονται και διαδίδονται πάρα πολύ γρήγορα στο ίντερνετ και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους παραγωγούς ε, ή το προϊόν. Αλλά η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτές τις ατομικές γνώμες με νομοθεσία, χωρίς να λάβει υπόψη και χωρίς να καταπιέσει και να παρεμποδίσει την ελεύθερη έκφραση άποψης. Επίσης η έκθεση μιλάει για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Θετικό αυτό και για τις διεθνείς προς τα παιδιά. Η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές επίσης το αναφέρει αυτό το θέμα. Όπως λέει η έκθεση, η Κομισιόν θα εξετάσει την εμπειρία των κρατών μελών από την οδηγία όταν ε, ετοιμάσει την έκθεση που αναμένεται το 2011 για την οδηγία. Την εμπειρία, την εμπειρία των κρατών μελών θα τη λάβουμε υπόψη μας στην έκθεση που ετοιμάσουμε, όπως είπα, το 2011. Είναι σημαντικές αυτές οι εμπειρίες για μας των εθνικών αρχών. Απατώντας τώρα στην ερώτηση της κυρίας Στήλερ, για το πλυντήριο. Μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική διαφήμιση με βάση την οδηγία της αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αν ένας, ας πούμε, εμπορευόμενος παρουσιάσει ως κάτι παραπάνω, ως κάτι ιδιαίτερο, ας μια προστιθέμενη αξία, την υποχρέωση, ας πούμε, που έχει ούτως ή άλλως με βάση την νομοθεσία στα πλαίσια της εγγύησης να δώσει αυτές τις δυνατότητες. Και αυτό αναφέρεται στο, ε, στο σημείο 10 του παραρτήματος ε, της οδηγίας. Ε, το καλύπτει αυτό το θέμα του πλυντηρίου η νομοθεσία μας. Λοιπόν. Ο κύριος Μπούντερ από την Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία των Πληροφοριών θέλει να πει και αυτός κάτι, αν το επιτρέπετε. Παρακαλώ. Η έκθεση αναφέρεται σε πολλά σημεία στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Να σας υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ε, δημοσίευσε την ε, ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη που περιλαμβάνει και τις ε, διαδικτυακές υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και παρόλο ότι δεν αναφέρεται ρητά στην διαφήμιση μέσω διαδικτύου η ψηφιακή ατζέντα έχει στοιχεία τα οποία είναι σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ένα από αυτά είναι ότι αναγνωρίζει την ανάγκη να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή έτσι ώστε να ε, καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την έλλειψη πίστης του καταναλωτή, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω, διαδικτύου. Ε, Επίσης ε, θέλαμε ε, να δημιουργήσουμε ένα κώδικα δικαιωμάτων ε, στο διαδίκτυο, στα οποία δικαιώματα ο καταναλωτή να βρίσκει απαντήσει απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Μια άλλη δραστηριότητα προβλέπεται είναι ε, δημιουργία μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων και φορέων ε, εμπλεκομένων φορέων για μια ειδική σήμανση αξιοπιστίας στις ε, ε, πωλήσει μέσω διαδικτύου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί η έκθεση αυτή είναι πολύ ισορροπημένη. Αναφέρεται στην έκθεσή του και, γιατί, και στην οδηγία ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών την γνωστή AVS οδηγία, η οποία επίσης διαθέτει διατάξεις για την προστασία καταναλωτών, ανηλίκων για παράδειγμα, ε, προστασία τους έναντι υπερβολικής ε, ε, διαφήμισης. Η Κομισιόν θα ενημερώσει μέχρι το τέλος 2011 για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και θα αξιολογήσει και το θέμα της διαφήμισης ε, στην τηλεόραση και ιδιαίτερως μέσω παιδικών προγραμμάτων. Θα αξιολογήσουμε επίσης και τη, θα λάβουμε υπόψη επίσης και τη δική σας έκθεση που συζητάτε σήμερα. Ε, έγινε, γίνονται λόγο στην έκθεση και για ε, ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, θέματα απορρίτου προσωπικών δεδομένων κλπ. Όλα αυτά ρυθμίζονται στην ε, οδηγία ε, προσωπικών δεδομένων, την οδηγία privacy και εκεί υπάρχουν διατάξεις βέβαια που επιτρέπουν στους ε, χρήστες να με ένα απλό τρόπο να αρνούνται εκ των προτέρων να λαμβάνουν ε, διαφημίσεις από εταιρείε κλπ. Η λήψη των διαφημίσεων πρέπει να γίνεται ε, μετά από ρητή συγκατάθεση. Να σας υπενθυμίσω τις καινούριες υπηρεσίε μέσω του διαδικτύου, οι οποίες χρηματοδοτούνται πολύ συχνά από έσοδα που προέρχονται από διαφημίσεις ε, μέσω διαδικτύου. Συνεπώς, ας μην υποτιμούμε την σημασία της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Στόχος της Κομισιόν είναι να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη αυτών των διαδικτυακών υπηρεσιών ε, δεν θα υποσκαφθεί και ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται απρόσκοπτα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζουβά για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Η ώρα προχωράει, θα είμαι λακωνικός. Συνολικά συμφωνώ με τις παρατηρήσεις. Ε, ε, ε, το ευάλωτο διαφόρων κατηγοριών, η αυτορύθμιση, η συρρύθμιση, το θέμα ε, το, του κοινωνικού και ψυχολογικού στοιχείου, της διαφήμισης που είναι πολύ σημαντικά, η έννοια... Αυτά που είπατε για, τα, για κάποια ειδικά προϊόντα, καπνό, αλκοόλ, φάρμακα, τα φάρμακα είναι τελείως διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Το, τα καπνά και το αλκοόλ αρχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει μια νομοθεσία για τα φάρμακα και δεν θα πρέπει να υπάρξουν τώρα επικαλύψεις, να μην κάνουμε και άλλα πράγματα σε αυτά που υπάρχουν. Επίσης, τη διαφήμιση τη ζουν διαφορετικά τα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, συχνά όταν κάνουμε ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε διαφημίσεις, α, μια διαφήμιση ας πούμε και τη συγκρίνουμε την αντίστοιχη στη χώρα μας. Ε, μερικές φορές εκπλησόμεθα από τις διαφορετικές αντιδράσεις. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εθνικές διαφορές ε, και να θεωρήσουμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουν την ίδια διαφήμιση. Δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι αυτό ζητούμενο. Το θετικό είναι ότι το ζήτημα του πλυντηρίου καλύπτεται, έχει ρυθμιστεί. Τώρα μπορώ να λάβω λοιπόν τις ε, προτάσεις ε, ε, τροπολογιών σας, τις οποίες θα τις επεξεργαστώ μαζί με τους κοιόδης συζητητές από την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Φτάσαμε 28-29 Σεπτεμβρίου για τις 5 ε, Οκτωβρίου μάλλον για τις τροπολογίες, 26-27 ε, ψηφίζουμε στην ΙΜΚΟ και ψηφίζουμε στην Ολομέλεια την έκθεση ε, τον Νοέμβριο. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, έπρεπε να, τελειώ... να τελειώναμε στις 6. Έχουμε ήδη ένα τέταρτο καθυστέρηση. Το θέμα είναι η βελτίωση τη οικονομική διακυβέρνηση και του πλαισίου σταθερότητα τη Ένωση ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Αφήνω το λόγο στον κύριο Κορέι Αντεκάμπο για να παρουσιάσει το θέμα. Θα ήθελα συνοπτικά να υπογραμμίσω τη σημασία αυτής της ε, ανακοίνωσης της Επιτροπής επί της οποίας ε, γνωμοδοτούμε. Η ανακοίνωση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης αλλά έχει και δομική σημασία διότι θα επηρεάσει τα επόμενα, πολλά επόμενα χρόνια τις σχέσεις των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, δικές μας ζωές ως πολιτών. Ζητώ συγγνώμη Όποιο δεν ενδιαφέρεται για τη συζήτηση, α βγει έξω. Παρακαλώ, μη συζητά σε πηγαδάκια. Ε, ε, Τέλος, ε, είναι σημαντική αυτή η γνωμοδότηση και για τη δική μας Επιτροπή, μάλλον για την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς, διότι ε, μας δίνει την ευκαιρία να επαναλάβουμε και να τονίσουμε τις πάγιες θέσει μας. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή της Επιτροπής ΕΚΟΝ, τον κύριο Ντιόγκο Φέιο. Στις 12 Μαΐου συναντήκαμε μια πρώτη φορά ε, και χρειάστηκε να καθυστερήσουμε λίγο διότι η ανακοίνωση Επιτροπής ε, δεν ήταν πλήρης. Ζητώ συγγνώμη, ε, λίγη ησυχία, γιατί πρέπει να σεβαστούμε λίγο και τον εισηγητή. Σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βασιζόμαστε λοιπόν στο έγγραφο της ε, Κομισιόν της 12 η Μαΐου αλλά και στην επόμενη εκδοχή του εγγράφου της 30ης Ιουνίου. Συμφωνούμε εν γέννη με, τα 8, με τις οκτώ συστάσεις. Έχουμε κάποιες προτάσεις τροπολογίας προκειμένου να εστιάσουμε καλύτερα το βλέμμα μας στην σταθερότητα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ε, συμφωνούμε με την υποστήριξη της ε, ε, πράξης μενίας αγοράς και της έκθεσης Μάριο Μόντι. Λέμε ότι πέραν του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να υφίσταται και ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης. Ίσως κάποιος μπορεί να πει ότι είναι δύσκολη η ε, μέτρηση της απασχόλησης, αλλά έχουμε το, το έγγραφο Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 που μας δίνει το πλαίσιο μέτρησης της ανάπτυξης, αύξησης της απασχόλησης. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εδώ. Οι, ε, έχουμε δείκτες, οι δείκτες ε, που συνοδεύουν το Σύμβολο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να συνοδεύονται με τη σειρά τους από δείκτες για τη γενική οικονομία όπως αυτοί που αναφέρονται στο έγγραφο Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Ε, για παράδειγμα, δείκτες για την ε, έρευνα, δείκτες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δείκτες για την εξέλιξη της απασχόλησης, της ανεργίας, της φτώχειας κλπ. Με αυτόν τον ε, τρόπο θα λάβουμε καλύτερα υπόψη την κατάσταση σε κάθε κράτο μέλο. Δεν θέλουμε να λαμβάνονται αποφάσεις αυτομάτως από την Κομισιόν χωρίς έγκριση του Συμβουλίου. Ε, προβλέπουμε κίνητρα θετικά και αρνητικά, τα οποία όμως θα πρέπει σίγουρα να περνούν από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει και όχι η Κομισιόν να ερμηνεύει κατά το δοκούν και αυθαίρετα την συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζεται σύσταση για την ενίσχυση της γραμματείας και ε, ε, της γραμματείας του, του Eurogroup. Δεν νομίζουμε ότι είναι αυτός εδώ, αυτό το εδώ το κατάλληλο σημείο, το κατάλληλο κείμενο για να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε γρήγορα μια ευρωπαϊκή υπηρεσία χρέους ε, για την παροχή εγγυήσεων και τη μείωση της κερδοσκοπίας εις βάρος των κρατικών χρεών. Χρειάζεται επίσης να προβλέψουμε τη δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων ε, πραγματικών ευρωμολόγων που προτάθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα και από τον κύριο Μπαρόζο. Ε, ο κύριος Μπαρόζο μίλησε για, το, για ε, ομόλογα project, ευρωπαϊκών project που συνδέονται δηλαδή με συγκεκριμένα μεγάλα ευρωπαϊκά project. Χρειάζεται, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για το συντονισμό, το συντονισμό των φορολογικών πολιτικών και δημοσιονομικών προοπτικών. Άλλωστε αυτό προβλέπεται και από το Single Market Act ρητά. Μιλάει μάλιστα για την εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών εκεί πέρα, Single Market Act. Όχι μόνο για το συντονισμό. Υπάρχουν, σχέση, υπάρχουν όμως θέματα όπως το ε, εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία μας αφορούν ιδιαίτερα σε σχέση με την εναρμόνιση αυτής, των φορολογικών πολιτικών. Γι' αυτό το αναφέρουμε κι εμείς. Παρόλο που αναφέρεται και στη Single Market Act. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους σκιώδους που συνεργάστηκαν πολύ ε, παραγωγικά μαζί μου. Είμαι ανοιχτό. αν μπορέσουμε να πάμε ακόμη πιο μακριά, στις συμφωνίες οποίες έχουμε καταλήξει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Περιμένω τις προτάσεις τροπολογίας σας και είμαι πρόθυμος να ξαναγράψω μερικά ε, σημεία του κειμένου. Μέχρι τώρα ήμουν πολύ απασχολημένος, τώρα όμως έχω περισσότερο χρόνο ε, και θέλω να ακούσω την άποψή σας. Τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ που δείχνετε ανοιχτό πνεύμα. Έχουμε ένα ταρτάκι περίπου για τη διερμηνία. Γι' αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσουμε τη συνεδρίαση. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Στον κύριο Ζουβά. Τρεις παρεμβάσεις έκανε σήμερα, θα κάνει σήμερα. Αντικαθιστώντας κάποιον άλλον σκιώδη εισηγητή. Ευχαριστώ. ε, αντικαθιστώ τον κύριο Λεγκρίπ, που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Ε, υπάρχουν δύο μείζωνα θέματα που μας δημιουργούν ε, πρόβλημα. Καταρχάς το σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης. Προφανώς, σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, ανάπτυξης και απασχόλησης, πολύ δίκαια και σωστά τους αναφέρατε, αλλά μπορούμε να τους υλοποιήσουμε μόνο, την, ε, μόνο μέσω και χάρη στην εξυγίανση ε, των δημοσιονομικών μας και τη μείωση του χρέους. Ε, το, ένα επιπλέον σύμφωνο έχει, δεν νομίζετε ότι μπορεί να είναι πολύ δεσμευτικό για τις οικονομίες. Ε, δεν δημιουργούμε, δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που δεν είναι σωστό. Το δεύτερο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το χρέος που προτάθηκε. Στο ΕΛΚ έχουμε πολλά προβλήματα με αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει κίνδυνος εδώ. Γιατί τα δάνεια που θα γίνονται ε, θα έχουν όλο και χειρότερες ε, συνθήκες. Ε, γιατί θα μπουν μαζί όλες οι χώρες στο ίδιο καλάθι, χώρες που έχουν καλούς βαθμούς και χώρες που δεν έχουν καλούς βαθμούς. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό ταμείο, νομισματικό ευρωπαϊκό ταμείο για το σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τις χώρες της Ευρωζώνης με βάση το, τον πλούτο του, το ΑΕΠ του δηλαδή. και ανάλογα με τις ε, παρεκκλήσεις από τα κριτήρια ε, για το χρέος. Αυτά τα είπα πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος σκιώδης, συγητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ζιβέν, συμφωνώ με τις ε, αντιρρήσεις σας στο σχέδιο της Επιτροπής έκον ε, λείπουν κάποια πράγματα αλλά δεν ξέρω και με τις ε, συνεισφορές του συγητή τι γίνεται. Κοιτάξτε, με τους φιλελεύθερους δεν θα κάνετε κανένα βήμα προς ε, μια τέτοια ένωση την οποία θέλετε. Δηλαδή, θα πρέπει ίσως ε, να δούμε το τι θα γίνει με μία προγραμματισμένη ίσως ε, χρεοκοπία των κρατών μελών και να πάει ένα 60% πιθανώς σε ευρωομόλογα και το υπόλοιπο βεβαίως ε, θα το επομιστούν ηλικία του Κάλα. Τέλος πάντων δεν έχουμε φτάσει ποτέ εδώ πέρα. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία το κράτος, το κοινωνικό το χρηματοδοτούν από τους φόρους ενώ η Γερμανία, παραδείγματο χάρη, χρηματοδοτεί το κοινωνικό κράτο μέσω εισφορών. Τι θα αρμονιστεί από αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Εκτός αν μπορούσαμε στον φόρο των επιχειρήσεων να κάνουμε μια κοινή φορολογική βάση. Αυτό έχει κάποια πιθανότητα και είναι και κάπως σχετικό ε, απλό. Αλλά έχω πολύ μεγάλες αμφούλειες ε, για το εάν το θέλουν τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο προβλέπεται λοιπόν ως pooling δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα είναι άλλο ένα βήμα προς μία αναδιανεμητική ένωση, μια αναδιανεμητική ένωση την οποία σας το λέω ξεκάθαρα θα απορριφθεί διακομματικά στην Γερμανία και υπάρχουν οπωσδήποτε και άλλες χώρες οι οποίες θα κάνουν το ίδιο οπότε δεν θα υπάρξει καμία πλειοψηφία. Οπότε θα καταθέσουμε και τις αναλογές τροπολογίες ε, στην έκθεση του συγκητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος λόγω του χρόνου. Θεωρώ πως ε, όταν ε, έχουμε μια γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ έχουμε δύο βασικά έγγραφα, την έκθεση Γκρέκ και την έκθεση του καθηγητή Μόντι και οι δύο τόνισαν πως για να λειτουργήσει πραγματικά η εσωτερική αγορά στο μέλλον πρέπει να δούμε την κοινωνική πτυχή. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχω εγώ εδώ πέρα με τις ε, προτάσεις ε, που γίνονται εδώ πέρα, δηλαδή πράγματι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα ελλείμματα του προπολογισμού. Σε αυτό συμφωνούμε, δεν είναι δυνατόν να επομίζονται αυτά τα βάρτα. Κοινωνική πτυχή, την καταπολέμηση στόχιας κτλ. Οπότε χαιρόμαστε βέβαια για την προσοχή στην οποία, η οποία αποδίδεται σε αυτά τα ζητήματα, αλλά πρέπει να δούμε την εσωτερική αγορά που είναι η βάση και το πώς θα μπορέσουμε να την διευρύνουμε. Επίσης το πρόβλημα το οποίο έχουμε από την άλλη είναι πως ποιες είναι οι κυρώσεις όταν δεν... Ε, καθώς υπάρχουν κυρώσεις εάν δεν μειώσει κανείς το έλλειμμα του υπερπολογισμού, αλλά δεν υπάρχουν κυρώσεις για τη φτώχεια και την ανεργία. Τώρα για τα των φόρων συμφωνώ τελικά με τον ε, κύριο Κρότσμαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περίμενα την ε, διερμηνία. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις για το χρέος. το θέμα του χρέους που θα πρέπει να υπο... βασίζεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. And uh, Για την ευρύτερη δέσμη των δικτών και το σύμφωνο απασχόλησης. Βασικό είναι να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά θέματα, δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Αυτό ήταν προβληματικό μέχρι τούδε. Δεν πρέπει να έχουμε πληθώρα δικτών. Γιατί με πάρα πολλούς δείκτες μπορούμε να το, μπορεί και να το αποδυναμώσουμε το σύμφωνο παρά να το καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό. Έχουμε τη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου της Task Force ε, του Φανρόμπουη. Η Κομισιόν θα προτείνει το νομοθετικό της πακέτο στις 29 Σεπτεμβρίου που θα συζητηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ και θα συζητηθεί επίσης και στο, στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Αυτές είναι οι επόμενες βασικές προθεσμι... Ε, ημερομηνίες. Και τώρα, τα τελικά σχόλια από τον εισηγητή. Ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές για τα σχόλιά τους. Τα σημείωσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερος ε, αυτούς που διαφώνησαν μαζί μου ειλικρίνεια σε δύο-τρία σημεία. ε, υπάρχει πεδίο διαπραγμάτευσης. Δεν πιστεύω ότι η απασχόληση θα πρέπει να είναι εκτός των, ε, του, του επικέντρου ενός Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ούτε και υπάρχουν επιχειρήματα να, υπέρ του ότι η απασχόληση είναι, ότι η απασχόληση είναι ε, εξαρτημένη μεταβλητή. Ε, είναι και αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή όπως και οι υπόλοιπε και είναι δυνατόν να μετρηθεί. Μην ξεχνάμε το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το, ευρωπαϊκό, το κοινωνικό πρόσωπο ε, δεν μπορεί να επισκιάζεται από τις συνθήκες, από τις συγκύριες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το διατηρήσει. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρέους, είμαστε ανοιχτοί. Είμαι ανοιχτό. Θα μπορούσα να δεχτώ και άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Είναι θέμα τεχνικό, ε, περίπλοκο. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι η πιο αρμόδια να τοποθετηθεί επί τέτοιων θεμάτων. Πλην όμως ε, να σας πω ότι το δικό μου σημείο αφετηρίας ε, δεν είναι πλήρως ασυμβίβαστο με την πρόταση του κυρίου Ζουβά. Σε ό,τι αφορά την φορολογική εναρμόνιση δεν έχει νόημα να ξαναξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Είναι άκρος ιδεολογικό το ζήτημα, αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω μόνο ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Αν θέλουμε μια εσωτερική αγορά, θα πρέπει να διαθέτουμε μηχανισμούς που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της. Και γνωρίζουμε ότι η φορολογική ποικιλομορφή αυτή τη στιγμή αποτελεί βαρύδι στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, πολύ δε περισσότερο που αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε προς ε, μία από αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέρουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ ξανά μία ακόμα φορά, λέω, τους ε, ηγητές. Θα τα ξαναπώ μαζί τους για να προχωρήσουμε περισσότερο το κείμενο συνενετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για αύριο λίγη στις 14 Σεπτεμβρίου στις 12 ε, η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσουμε το κείμενο. Ε, θα ψηφίσουμε μάλλον και στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε ψηφίσουμε την έκθεση. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ.